I think we can start. Νομίζω... Δεν απατώμε, λέω να αρχίσουμε. καλωσορίζω και κυρίω την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης. Μπορεί να εγκριθεί η μερίσια διάταξη αν δεν διαφωνεί κανείς. Όπως και δεν διαφωνεί. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης 9 και 10 Νοεμβρίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ενστάσεις θεωρούνται τα πρακτικά εγκεκριμένα. Ανακοίνωση του Προέδρου. Δεν έχω καμία ανακοίνωση προς το παρόν. Συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τη διαπραγματεύση σχετικά με τη Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών. Η είναι ο κύριος Παντενκάμπ, είναι το θέμα της ΤΙΣΑ, δεν μιλάει κανείς, ψηφίζουμε μόνο. Η συζήτηση έχει γίνει, έλεγχο πρώτα, αν είστε όλοι παρόντες και έτοιμοι με τις κάρτες σας. Όλοι εντάξει είμαστε ούτε υπεράριθμους έχουμε μια χαρά. Πραγματικά έτσι μου φεύγει ένα βάρος. Λοιπόν, πάμε. Τροπολογία παριθμό 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία παριθμών 4 υπέρ. Κατά. άποχε, απορρίψετε. Η συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμών 10 υπέρ. Κατά. άποχε, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία μόνο 11 ψήφι πέ. Κατά. Άποχες έλεγχος παρακαλώ. Έχει την ψηφοφορία. Μια στιγμή να δούμε να ψηφίσουμε όλοι. Για να ψηφίσει και ο κύριος Δεγκράντες Πάσκουαλ. Τώρα ελπίζω να μην είναι ο υπεράριθμος. Πέρασε. Μάλιστα. Βέβαια, Ισμαήλ, εδώ έχουμε ίσα δικαιώματα όλοι. Και όλοι οι καθυστερημένοι επίσης. Paul, sag, sag, sag ihm. ihm. Εντάξει, το ελέγξαμε, έχουμε ακόμα περιθώριο, δεν περισσεύει κανείς. Jetzt um Είναι και δική του τροπολογία. Μπα, δική σου τροπολογία, γι' αυτό σε περιμέναμε. Και τώρα λέει Ισμαήλ τέρμα. Λοιπόν, ψηφίζουμε την τροπολογία 11 του Μπα Αικχάουτ. Πρέπει να βγάλει και την κάρτα του. Ωραία, είναι και έτοιμο. Πάμε. Πέρας. 19 ε, απορρίπτεται με μικρή διαφορά 19 υπέρ 21 κατά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τροπολογία 75. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Η 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, η τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές έλεγχος στην τροπολογία 55. Άρχιτε ψηφοφορία και λίγη τώρα. Απορρίπτεται 19 υπέρ, 23 κατά. Η συμβαστική 3 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 26 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τσεκ, με χαρά. 26 λοιπόν ελέγχουμε την τροπολογία. Αρχίζει τώρα. Πέρας. 22-20 εγκρίνεται. Με μικρή διαφορά είχατε δίκιο, ήθελε έλεγχο. Η τροπολογία με 25 ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 πέρα, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 34 ΕΠΕ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ στην 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται 17-25. 33 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό θέλει έλεγχο. Είμαστε στην 33. η ψηφοφορία. Πέρασε. Με μία ψήφο διαφορά. 21 υπέρ, 22 κατά. Απορρίπτεται. Η 32 ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος για την 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 19-23 απορρίπτεται. Η 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 30. Άχι την ψηφοφορία. Ορίστε. Πέρας. 20-18 εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Η τροπολογία 35 υπέρ. Όχι, όχι, καταπίπτει λάθος έκανα. Πού πάμε τότε. Στην 36 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 38 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται 15-24. Τροπολογία 40. Ε, Ψήφι Π. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Γιατί την 39 η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Το ίδιο 21. Τροπολογία παριθμών 22. καταπιπτει Καταπίπτει 22. Και πάμε σε 41. Ψηφιπέ. Κατά. Έλεγχος. Στη 41 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία απορρίψεται. Η 53 ψήφι πέρα. Κατά. Και αυτό έλεγχο, και αυτό. 53 ηλεκτρονικά αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Το αυτό, ισοψηφία απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Συμβαστική 4 πέ. Κάτω. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμό 47. Ψήφι πέ. Κατά. Έλεγχος. 47. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. 18-22. Απορρίψετε. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Γιατί 48. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία απορρίπτεται. 21-21. Η τροπολογία υπερθών 49 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Στην 51 αρχίζει ψηφοφορία. Τελειώνει. Απορρίπτεται 15-25. Η τροπολογία υπερθών 50, το δεύτερο τμήμα μόνο λέει εδώ, υπέρ, κατά, έλεγχος και πάλι για την 50, το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. 20-22 απορρίπτεται. Η τροπολογία παρθών 12. Υπέρ, κατά, άποχες, έλεγχος και αυτό. Στη 12. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 18-24 απορρίπτεται. Η 54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 65 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μόνο σου ήσουν από τη δική μου ομάδα δεν ψηφίζαν οι υπόλοιποι. Εγώ τι να κάνω τώρα. Έλεγχο θέλετε είμαστε εντάξει. Έλεγχος. Στην 67 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 64 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 68 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση γιατί είναι 68 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. 22-20 εγκρίνεται. Ναι, και εγώ δεν θα το έχω φανταστεί. Ε, συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 13 τώρα, επέρ. κατά, έλεγχος, στη 13, αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται 21-22. Η 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτή θέλει έλεγχο. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη. 19-20. Απορρίπτεται. Καλά. Τρελά πράγματα. Η 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και πάλι έλεγχος. Στην 57 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασα. Μία ψήφο διαφορά απορρίψετε. 21-22. 73 υπέρ. Κατά. Και αυτό θέλει έλεγχο. Στην 73 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. 20-22. Απορρίπτεται. Ή 74 Υπέρα. Κατά. Άποχες. Απορρίψετε. Ή 76 Υπέρα κατά αποχές έλεγχος για την 76 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας 15-23 απορρίπτεται η τροπολογία 27 ψήφι πέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 ε, πέρα, κατά αποχές έλεγχος στην 56 αρχίζει ψηφοφορία. Περάστε. 20-22 απορρίπτεται. Η τροπολογία 78 ψήφι Κατά. Άποχες, έλεγχος και γι' αυτό στην 78. Αρχίζει ψηφοφορία. Περάστε. 18-22 απορρίπτεται. Η 79 υπέρ. Κατά. Αποχές, έλεγχος και πάλι την 79 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. 22-21 εγκρίνεται με μια ψήφο διαφορά. Η τροπολογία υπέρθμων 80 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Στην 80. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. 22-21. Δεν κρίνεται. Τροπολογία υπαριθμό 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία υπαριθμών 1. Διολογικές σκέψεις υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τσεκ. Καλά. Την τροπολογία υπαριθμών 1. Λοιπόν, τσεκάρουμε. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται η ισοψηφία 21-21. 21-21 ισοψηφία απορρίπτεται. Και μία αποχή ήταν. Η τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Τσεκ. Στη 2. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 20-22. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα. Περιμένουμε λίγο. Άλλοι τρεις να ψηφίσουν παρακαλώ. Τώρα λίγοι. 27, 14 και μία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά μου, Βίμ Φαντεκάμπ. Ja. Also solche knappen Abstimmungen, Τόσες πολλές ε, ψηφοφορίες με τόσο μικρές διαφορές ε, σπάνια είχαμε στην Επιτροπή μας. Πάμε. Στο επόμενο θέμα λοιπόν, υπαριθμό 5 παρουσίαση από την Επιτροπή ενός μέτρου επιτροπολογίας σχετικά με την ταξινόμηση σοβαρών παραβάσεων στις οδικές μεταφορές. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για μια πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ταξινόμηση παραβάσεων στις οδικές μεταφορές που μπορούν να οδηγήσουν στην αφαίρεση της άδειας ε, λειτουργίας σε μεταφορικές εταιρείες αν δεν βάλει βέτο μέσα σε τρει μήνε στο Κοινοβούλιο, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε αυτό το μέτρο. Βιμ Βαντενκάμπ. Όπω γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρυσι ε, επανέπεψε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετική πρότασή της και στη συνέχεια την επεξεργάστηκε και την καταθέτει ξανά προς έλεγχο στο Κοινοβούλιο και εξέταση για να μπορούμε να ασκήσουμε κανονικά ε, το καθήκον μας και ε, να αποφασίσουμε με τα λόγου γνώσεως παρακάλεσα τη Γενική Διεύθυνση MOVE να έρθει να μας τα παρουσιάσει σήμερα στην Επιτροπή μας. Έχετε το λόγο λοιπόν κύριε Λιζουά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλή σας σήμερα. Το Κοινοβούλιο έλαβε μία νέα έκδοση της ταξινόμησης των σοβαρών παραβιάσεων που πρόσφατα ψηφίστηκε στις 13 Οκτωβρίου από την Επιτροπή Μεταφορών η προηγούμενη εκδοχή υπευλήθη στο Κοινοβούλιο πριν από ένα χρόνο, αλλά περίφθη από το Κοινοβούλιο βασικά για δύο λόγους. Πρώτον, ότι το Κοινοβούλιο θεώλησε ότι ορισμένες παραβάσεις δεν ορίζονται σαφώς και άλλος λόγος ήταν ότι σύμφωνα με το Κοινοβούλιο ότι έλειπαν πολλές παραβάσεις και δεν υπήρχε συμμόρφωση με τους κανόνες του Καμποτάζα. Η Επιτροπή επανασυνέταξε μία εκδοχή που βεβλίδη στο Κοινοβούλιο. Τονίζω και πάλι ότι αυτή αναδιαμορφώθηκε από κοινού με 28 εθνικούς εμπειρογνώμονες. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές αρχές ελέγχου, από τις χώρες μέλη. Ήταν συνεπώς πολύ σημαντικό για την Επιτροπή να ψηφιστούν τα μέτρα από τις χώρες μέλη, όχι απλά με πλειοψηφία, αλλά με μια πολύ μεγάλη στήριξη. Θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να υιοθετηθούν τα μέτρα αυτά. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι βασική η προτεραιότητα να υπάρχει ενιαία εφαρμογή της νέας νομοθεσίας. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε και μία ενιαία ταξινόμηση των σοβαρών παραβάσεων που θα αποτελέσουν ένα κοινό σημείο αναφορά για να γίνει μία αξιολόγηση των διαφόρων φορέων και αυτό θα επιτρέψει και στις χώρες μέλη να ανταλλάξουν πληροφορίες για το σύστημα ΕΡΟΥ, δηλαδή το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης. Τι κάναμε Ουσιαστικά λάβαμε υπόψη μας τις παρατηρήσεις και τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο πριν από ένα χρόνο. Πρωτίστως προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε στο μέτρο του δυνατού τον ορισμό των παραβάσεων και να γίνει σαφέστερος Τονίζω ιδιαίτερα τις παραβάσεις που αφορούν την εξαίρεση των 12 ημερών ε, αλλά και το, τα πιστοποιητικά που αφορούν τους οδηγούς. Λάβαμε υπόψη σας και την ευκαιρία της αναθεώρησης του πρώτου σχεδίου κανονισμού για να συμπεριλάβουμε και άλλες παραβάσεις. Μη συμμόρφωση, για παράδειγμα, με την ε, περίοδο οδήγησης πριν να υπάρχει ένα διάστημα ε, ανάπαυσης ή το θέμα που αφορά τον ταχογράφο. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μία συγκεκριμένη παράβαση που αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών. Φροντίσαμε έτσι ώστε οι παραβάσεις που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο είναι ε, ε για τα οποία θα θεωρείται υπεύθυνος ο μεταφορέας και όχι ο αποστολέας. Η ευθύνη λοιπόν αφορά το μεταφορέα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επέκταση του καταλόγου των παραβάσεων σε άλλες παραβάσεις και ιδιαίτερα στην παράβαση της μη συμμόρφωσης με τους κανόνες του, ε, της ακτοπλοείας. Το καμποτάζ δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο που έχετε μπροστά σας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το, η παρούσα εντολή που έχουμε να καταρτήσουμε αυτό το κατάλογο παραβάσεων δεν αφήνει περιθώρια να συμπεριληφθεί το παράνομο καμποτάζ από τη στιγμή που οι παραβάσεις θα πρέπει να ε, άπτονται της οδικής ασφάλειας. Θα έλεγα ότι ε, η συμπερίληψη αυτό είναι το πρώτο βήμα, το δεύτερο είναι να ταξινομηθούν οι παραβάσεις, οι παραβάσεις ε, ε, που είναι και τη σοβαρότητα των παραφάσεων και θέλουμε να συμπεριλάβουμε το παράνομο καμποτάζ, αυτή η παράβαση θα θεωρηθεί παράβαση ελάσσονος σημασίας, θεωρώντας την επίπτωση που έχει στην οδική ασφάλεια. Όλοι γνωρίζετε βεβαίως ότι η Επιτροπή επεξεργάζεται μία πρωτοβουλία για θέματα οδικής ασφάλειας που θα υποβληθούν στο τέλος του 2016 ε, ε, και πρόθεση της Επιτροπής είναι να προτείνει ως μέρος μίας αναθεώρησης του βασικού κανονισμού 1071 του 9 μία επέκταση εντολής της Επιτροπής έτσι ώστε η Επιτροπή να μπορεί στο μέλλον να προτείνει έναν εκτενή κατάλογο παραβάσεων που θα συμπεριλαμβάνει και τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες του καποτάζ και να μπορεί να ταξινομεί τις παραβάσεις ανάλογα με την σοβαρότητά τους και αυτό θα βατισίζεται στην, στο, κατά πόσον επηρεάζουν τον ανταγωνισμό και τον υγιή ε, ανταγωνισμό αλλά και την ε, παραβίαση ε, άλλων κανόνων στους καταλόγους. Αυτά είναι τα βασικά σημεία επί των οποίων θα ήθελα να επιμείνω. Βεβαίως η Επιτροπή είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο ερώτημα σε μια μετέπειτα φάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Βίμ Φαντεκάμπ έχει πρώτο το λόγο ή δεν θέλεις. Καλά, ο Μάρκος Φέρμπερ τότε. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε στα αιτήματα του Κοινοβουλίου που εκφράσαμε τον περασμένο Δεκέμβριο στην Ολομέλεια και που τα πήρε και σοβαρά υπόψη γιατί αυτή την, πρόφαση, πρόθεση είχαμε, για να το πω ξεκάθαρα, σε πολλά σημεία υπάρχουν και διευκρινήσεις και βελτιώσεις για την εσωτερική ναυσιπλοεία είχα την ευκαιρία να συζητήσω με την αρμόδια επίτροπο για τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται επικίνδυνα υλικά στις ε, οδικές μεταφορές ε, και τις διεθνείς συμβάσεις. Θα πρέπει και αυτά να συμπεριλαμβάνονται. Ή άλλο θέμα, να έχουμε περισσότερη οδική ασφάλεια. Στη δική μας πολιτική ομάδα δεν το έχουμε ε, ολοκληρώσει αυτό το θέμα συζήτηση. Πάντω χαιρόμαστε που ανταποκρίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λαμβάνει υπόψη τη τα μελήματα και τι επιθυμίε του Κοινοβουλίου. Στην πρότασή τη τώρα θα μελετήσουμε το θέμα προσεκτικά, αλλά εκ πρώτη όψεω από ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτά που στο μεταξύ έχει φέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο Ισμαήλ Ερτούκ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και από τις δικής μας πλευράς της Σοσιαλιστών και Δημοκρατών την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ε, συμπεριέλαβε τα δικά μας μελήματα και εν μέρη τα έχει ε, υλοποιήσει. Εμείς οι σοσιαλιστές δεν μπορούμε να είμαστε 100% ικανοποιημένοι, παρόλα αυτά θα συμφωνήσουμε και θα υπερψηφίσουμε. Να σας πω τα θετικά. Πρώτον, η συμπερίληψη ε, του κανόνα λεγόμενου του 12 ημέρου και ε, η συμπερίληψη διαφόρων εγγράφων και ε, φορτωτικών και η χρήση ε, ταχογράφου που δεν είναι πιστοποιημένος ή εγκεκριμένος από αρμόδιο οργανισμό. Για όλα αυτά τα θετικά ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, από πλευράς εργαζομένων υπάρχουν ακόμα κάποιες ελλείψεις, το είπατε και εσείς ο ίδιος το παράνομο καμποτάζ δεν ελήφθη υπόψη. Και παρόλα αυτά εμείς θα συμφωνήσουμε και θα υπερψηφίσουμε για το λόγο και το λέω ξεκάθαρα ότι μας έδωσαν διαβεβαιώσεις ότι του χρόνου θα τα λάβετε υπόψη στο πακέτο στη δέσμη μέτρο για τις οδικές μεταφορές. Ε, είναι ψήφος εμπιστοσύνης αυτή των σοσιαλιστών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δίνουμε. Äh, ε, ε, τι άλλο θα πρέπει να διευκρινίσουμε. Εάν συζητήσουμε αυτό το θέμα του χρόνου και όταν το κάνουμε αυτό παρακαλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιλέξει σαφείς διατυπώσεις για να μην υπάρχει χώρος για παρερμηνίες. Αυτό το καιρό ας πούμε δεν είναι ξεκάθαρο. Τι σημαίνει, όταν πρόκειται για διαδικασία αφαίρεσης της άδεια λειτουργίας μιας μεταφορικής εταιρείας, ποιος χάνει ε, την άδεια εκείνος που έχει πάρει την ανάθεση, εκείνος που έχει δώσει την ανάθεση. Ο υπεργολάβος τρόπον την ή ο εργολάβος του έργου της μεταφοράς. Ε, και ε, σε περίπτωση ε, υποχρεωτικής τεκμηρίωσης με έγγραφα και παραστατικά επίσης θέλουμε σαφείς ορισμούς, θα συμφωνήσουμε και εμπιστευόμαστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του χρόνου όταν θα ξαναδεί την οδηγία 1071 το 2009 θα τα συμπεριλάβει αυτά. Ευχαριστώ, Ρόμπερτ Ζήλ. Uh, θα ήθελα να πω και εγώ με τη σειρά μου, ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από ένα χρόνο υποβάλλατε μια καινούρια ε, εκδοχή που αφορά τις παραβάσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε σοβαροί ως Κοινοβούλιο. τα σχόλια της Επιτροπής ε, ήταν ε, σαφή. Δεν υπά... Οι περιορισμοί δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την πρόταση. Το νομικό καμποτάζ είναι μία εντελώ ε, καινούρια... Το παράνομο καμποτάζ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και είναι ένας κίνδυνος όταν μιλάμε για την νέα αγορά. Βεβαίως δεν είμαι οραματιστής, Πιστεύω όμως ότι από την πολιτική άποψη θα πρέπει να σκεφτούμε τον τομέα των μεταφορών και να συμπεριλάβουμε στις οδοτικές μεταφορές κάτι που λέγεται ενιαία αγορά. Βεβαίως είμαι υπέρ, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και μερικές λεπτομέρειες ακόμα. Ευχαριστώ. Κι Στέλλα. Κι Δεν θέλω. Ο Κι Ναι. Ευχαριστώ. Βεβαίω ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το κείμενο της Επιτροπής είναι βελτιωμένο. Αλλά το καμποτάζ παραμένει ακόμα να καθόδες σημείο. Η ενιαία αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει από τη στιγμή που υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εργαζομένων. Το κοινωνικό ντάμπινγκ και ο θέμικος ανταγωνισμός είναι προβλήματα και είναι δική μας ευθύνη να τα καταπολεμήσουμε εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τομέας των μεταφορών πλήττεται από το κοινωνικό και αυτό έχει επιπτώσεις σε επίπεδο οδικής ασφάλειας. Επιπτώσεις που δεν είναι λάσονο σημασίας σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκλέγεται με καθολική άμεση ψηφοφορία έχει ένα σημαντικό ρόλο για να διαδραματίσει. Θα πρέπει λοιπόν να μην χαλαρώσετε τις προσπάθειές σας για το παράνομο καμποτάζ, παράλληλα όμως θα πρέπει να ενθαρρύνουμε όλες τις πρωτοβουλίες που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς μια επικοδομητική κατεύθυνση. Θα μπορούν να γίνουν πάρα πολλά έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο πλαίσιο. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό φορέα οδικών μεταφορών που θα μα επιτρέψει να εφαρμοστούν οι υπάρχουσε νομοθεσίες. Έχουμε κανονιστικά κείμενα που είναι καλά, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μεγαλύτερο έλεγχο τη εφαρμογή του, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή του. Γι' αυτό το λόγο με την ευκαιρία αυτή της ε, ε, κατεξουσιοδότηση πράξη, Θα παρακαλούσα την Επιτροπή να φροντίσει έτσι ώστε να εφαρμοστούν όλα αυτά τα κείμενα. Ευχαριστώ πολύ ο Πέτερ Λόντγκριν. Η να πω, τι Μα δεν καταλαβαίνετε πώς δουλεύουν οι μηχανισμοί της αγοράς και των τα αποτελέσματα της νομοθεσίας. Τι θέλετε ακριβώς. Να μας καταστρέψει ο ανταγωνισμός ή να ακολουθήσουμε τους κανόνες. Εδώ χρησιμοποιούνται οδηγοί με ξένες ε, άδειες οδήγησης σε τρίτων χωρών δηλαδή και οι οποίοι παρακάμπτουν την νομοθεσία. Το πρόβλημα με το καμποτάζ είναι ότι είναι πολύ εύκολο να υπάρξουν απάτες γύρω από αυτό. Από τη Σουηδία στη Δανία χρειάζονται 20 λεπτά με τη γέφυρα. Ξεφορτώνουν στην Κοπενχάγη και επιστρέφουν και μετά αρχίζει νέα περίοδος καμποτάζ όλα από την αρχή. Υπάρχουν συστηματικές απάτες η νομοθεσία για το καμποτάζ είναι από τις χειρότερες σε ολόκληρη την Ένωση γιατί επαναλαμβάνω είναι πολύ εύκολο να παρακαμφθεί. Στην αρχή υπήρχαν άδειε για επταήμερη οδήγηση και τώρα υπάρχει πλήρη απελευθέρωση ώστε να μπορεί κανείς να κάνει όσες όσα δρομολόγια θέλει. Εδώ χρειάζεται πολιτική απόφαση από το Συμβούλιο Υπουργών εκτός, από τον, εκτός ελέγχου της Κομισιόν. Ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους, πόσες απάτες και πόσες εταιρείες πλήττονται από αθέμητο ανταγωνισμό με οδηγούς που σχεδόν δεν έχουν άδεια οδήγησης. είναι σχεδόν αδύνατο η αστυνομία να ελέγξει τι ακριβώς συμβαίνει. Το πρόβλημα είναι ότι θέλουν οι οδηγοί να δουλέψουν όπως πρέπει αλλά δεν το καταφέρνουν. Και εσείς τα επιτρέπετε όλα αυτά. Ευχαριστώ χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή της. Λέει η κυρία Κράσβαντερ Χάιντς. Δυστυχώς δεν με ικανοποιεί η παρούσα πρόταση και στην Αυστρία διαφώνησε και το Συμβούλιο. Και θέλω να πω και για ποιους λόγους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρουσίασή της μας είπε ότι θα ληφθούν υπόψη μόνο οι παραβάσεις αυτές που είναι σοβαρές και μπορούν να οδηγήσουν σε ε, απώλεια ανθρώπινης ζωής. Μα ε, υπάρχει ο κανονισμός 1071 του 2009 που δεν τηρείται. Σύμφωνα με τις αιτιολογικές σκέψεις του λόγου κανονισμού ε, σκοπός είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αλλά και η εξασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού, βελτίωση της διαφάνειας στην αγορά, καλύτερη κοινωνική προστασία και ε, επίτευξη κοινών στόχων ε, και προτύπων. Με αυστηρά κριτήρια για την αξιοπιστία. Η επιχειρηματολογία που λέει ότι οι απαιτήσει του Κοινοβουλίου να συμπεριληφθούν και άλλα δικήματα όπως το παράνομο ε, και το κοινωνικό ντάμπινγκ επειδή δεν υπάρχει λέει η εντολή κατά την άποψή μου δεν ευσταθούν τα επιχειρήματα αυτά. Ε, από την άλλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπερεύει τις αρμοδιότητές της ε, όταν ε, βάζει νέα κριτήρια ανοχής όπως στα μέτρα και σταθμά, νέες κατηγορίες στην ταξινόμηση για ε, χρόνου οδήγησης και ξεκούρασης και ανάπαυσης. Και de facto αλλάζει ε, την κείμενη νομοθεσία. Επίσης υπάρχει και αρχή της αναλογικότητας την οποία παραβιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί οι παραβάσεις και η ταξινόμηση είναι τόσο περίπλοκες ε, και αντιτίθεται σε κείμενη νομοθεσία, σε οδηγίες και κανονισμούς και είναι νεφέλωμα ε, που δεν μπορεί κανείς να ελέγξει. Γι' αυτό θα παρακαλούσα την πρόταση όπως έχει σήμερα να την απορρίψουμε και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Πέτερ Φαντάλεν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Περί τίνος πρόκειται εδώ. Είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα ακρογωνίως λήθος τη ε, Ευρωπαϊκή πολιτική. Ε, Εμεί είμαστε πάρα πολύ καλοί στην έκδοση τη νομοθεσία, ε, κανονισμού και οδηγίε, αλλά η υλοποίηση και η εφαρμογή είναι ένα σημείο όπου χωλαίνει τα μάλα η πολιτική μα. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση λοιπόν στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάνω από ένα χρόνο ασχολούμαι προσωπικά και προσπαθώ να πάρω απάντηση από την Ευρωπόλ για τη πλαστογραφία ε, διαφόρων εγγράφων, φορτωτικών και τα λοιπά ε, και παραστατικών. Η Ευρωπόλ ε, δεν μου απαντάει, είναι απρόθυμη. Μπορεί να με φωτίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται με τη συγκεκριμένη πρόταση και με τις απάτες που γίνονται με πλαστογραφίες για φορτωτικές και ακόμα για διπλώματα οδήγησης και ποιες είναι οι ποινές και οι κυρώσεις που επιβάλλονται. Και πέρα από την ε, συγκεκριμένη ερώτηση έχω μια παρατήρηση. Με μεγάλη λύπη ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του 2016 θέλει να φέρει ε, μία πρόταση για τις οδικές μεταφορές. Ωραία αυτά που λέει ο κύριος Σερτούκο ότι τις δίνουν προκαταβολικά ψήφο εμπιστοσύνη, αλλά ε, να καθυστερήσει τόσο πολύ το πακέτο για τις οδικές μεταφορές θα μας πάρει άλλο ένα χρόνο. Και μάλιστα λέει ένα χρόνο πιθανώ. Χαιρετίσματα σου λέει πιθανώς ένα χρόνο κατάλαβε. Και το Team Juncker που είναι η σούπερ ομάδα και θέλει να προχωρήσει και να προωθήσει την Ευρώπη ε, σε τέτοια σημαντικά θέματα όπω είναι οι οδικέ μεταφορέ ε, θα πρέπει να περιμένει ένα χρόνο ίσως και παραπάνω. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κρίμα και θα ήθελα να ακούσω την ε, απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ο Μπρινό Ευχαριστώ Πρόεδρε, ομολογώ ότι αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Μάλλον θα έχω χάσει κάποιο επεισόδιο από την ταινία αυτή. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση για να αποβαθώ επί ενός κειμένου που ομολογώ ότι δεν γνωρίζω. Ίσως, ε, σίγουρα θα ήταν στην σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάντως ε, στα δικά μας έγγραφα εργασίες εγώ δεν τη βρήκα. Ε, και αυτό είναι ενοχλητικό. Πώς να αποφανθείς. Ε, δεν ξέρω, μπορεί να φταίω εγώ απολύτως, δεν, δεν ε, ρίχνω το φταίξιμο σε κανένα. δεύτερο, με πείθει πάρα πολύ αυτά που είπε κατηγορηματικά ο συνάδελφος Λούντρεγ με βρίσκουν σύμφωνο. Έχει δίκιο. Από την άλλη είμαι σε κάποια σύγχυση ε, για την έννοια αυτού του κανονισμού την ίδια. Δηλαδή τίνει να επιτρέψει την αφαίρεση άδειας λειτουργίας εταιρεία. Αυτό είναι εξαιρετικά βαρύ για τις εν λόγω επιχειρήσεις και έχει ποινικό χαρακτήρα. Και προβληματίζομαι. Διερωτώ με έχουμε εμείς τέτοια αρμοδιότητα. Να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις, τέτοιες φύσεως που έχουν να κάνουν με ποινικό δίκαιο. συνάδει πάρα πολύ με την αρχή της επικουρικότητας. Αυτή είναι μια επιφύλαξη που διατυπώνω και πάλι χωρίς να έχω διαβάσει το κείμενο. Επιφυλάσσομαι να αποκρισταλώσω οριστική άποψη όταν θα γνωρίζω περισσότερο για το θέμα. Ενημερωτικά θα ήθελα να πω ότι και εμείς μόλις χτες πήραμε το έγγραφο. Το στείλαμε όμως με το newsletter. Υπάρχει ένα σύνδεσμο, ένα link αλλά η αποφασιστική ψηφοφορία δεν είναι τώρα, είναι το Γενάρη. Έχετε αρκετό χρόνο να το διαβάσετε, να το μελετήσετε με την ισχύ σας και να διαμορφώσετε και άποψη. Τώρα έχει το λόγο Τζάκι Φώστερ. Ευχαριστώ. Δεν το είδα το έγγραφο χθε. Δεν το βρήκα δηλαδή. Θα ήταν όμως βοηθητικό γιατί όλους πάντα παίρνουμε τόσα πολλά έγγραφα να είχαμε το πρωί μια μικρή ενημεροσούλα τυπωμένη για να βρούμε ποια είναι τα συγκεκριμένα σημεία και τα συγκεκριμένα έγγραφα για να μην χρειάζεται να τα ψάχνουμε όλα. Θα μας, μας βοηθούσε πολύ. Τώρα για τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν νομοθεσία ήδη υπάρχουσα και εγχώρια από τα τοπικά κοινοβούλια και ενωσιακά. Αυτά που είπε ο Πίτερ τα καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τα σύνορα, το ξέρουμε αυτό. Αν δεν ελέγχονται στα σύνορα οι διακινήσεις, τότε είναι σχεδόν αδύνατο να βρούμε τη λύση. Λέμε, μιλάμε για απάτες, αλλά δεν είναι πάντα απάτες, είναι λυπής έλεγχος. Και υπάρχει και το εξής. Η διαφορά των νομικών συστημάτων και η ευθύνη ημί των οδηγών σε μερικές χώρες μέλη θα διωχθεί η εταιρεία ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο ο οδηγός. Πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Δεν θα αλλάξουμε όλα τα νομικά συστήματα όλων των χωρών. Τι θα χρειαστούν δεκαετίες. Αλλά να το δούμε λιγάκι αυτό και να λάβουμε υπόψη μας τις διαφορές και φυσικά ευχαριστώ και την Κομισιόν για την προσέλευσή της εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Για να το διευκρινίσω, η προθεσμία για τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις είναι στις 14 Ιανουαρίου, ενώ για την Ολομέλεια 28 Φεβρουαρίου. Έχουμε χρόνο να το κοιτάξουμε. Αλλά επειδή θέλαμε να γίνει μια συζήτηση, καλέσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρούσαμε ότι θα γίνει προφορικό αυτό. Ε, μας στείλαν όμως κείμενο και μόλις το λάβαμε, το στείλαμε και στους συντονιστές και στο newsletter. Ε, κύριε Σπαμίτλεμπορκ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Πρώτον, είναι καλή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τουλάχιστον για τις οδικές μεταφορές όπως και ε, η κυρία Φώστερ και ο κύριος Φαντάλεν, θέλω να πω ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται πάρα πολύ σωστά η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όχι μόνο με ενιαίο τρόπο και ε, ομοιόμορφο και στα 28 κράτη-μέλη, αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα ελέγχων και η διοικητική δυνατότητα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θα κάνει, ε, θα το ελέγξει αυτό, θα το παρακολουθεί. Είναι πολύ σημαντικό. Ο Επίτροπος Τίμερμανς έχει μια ατζέντα για εφνομοθετή. Καλύτερη νομοθεσία, better regulation το λένε. Καμιά φορά αυτό σημαίνει και λιγότερη νομοθεσία και λιγότερες φιλοδοξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πολλά πράγματα έχουν ε, οδηγηθεί σε εμπλοκή, έχουν φρενάρει. Περιμένουμε τόσο καιρό το πακέτο για τις οδικές μεταφορές και δεν ισχύουν τα επιχειρήματα αυτά που ακούμε. Ε, δεν είναι ε, ένα πακέτο, δεν είναι δέσμη νομοθετικό, από ό,τι ακούω είναι κατακαιρματισμένα. Και η Επίτροπος Μπούλτ θα φέρει κάποιες προτάσεις και είναι πακέτο, αυτό είναι δέσμη ή είναι νομοθετήματα δεξιά και αριστερά. Παρακαλώ να τα κοιτάξετε αυτά σοβαρά ε, και να είναι σαφείς οι κανόνες που διέπουν τις ε, μεταφορές, γιατί πραγματικά το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη μεταφορές στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και χειροκροτεί και ο Πέτερ Φαντάλιν που τον επενέσατε. Ο Ντομινίκ Ρικέ. Ευχαριστώ. Ας μην επαναλάβω ό,τι είπαν άλλοι. Είπαμε η Κομισιόν να ξαναδεί το θέμα του καμποτάζ αν και ίσως δεν είναι καταλληλότερο βήμα το κοινοβούλιο. Πάντως μερικές άλλες φορές που το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν κάποια αντίδραση υπήρξε. Τώρα τέθηκαν θέματα από τη συνάδελφο Λούντγκριν, τουλάχιστον για τα σοβαρότερα προβλήματα Δεν παραλαμβάνω όλα αυτά. Απλώς θέλω να τονίσω κάτι που μου φάνηκε περίεργο. Στον δεύτερο πίνακα για τις παραβιάσεις των ταχογράφων. Η Κομισιόν προτείνει για μερικές παραβιάσεις να θεωρήσουμε ποιες είναι οι σοβαρότερες. Serious infringement. Όταν κανείς αρνείται τον έλεγχο δεν είναι αυτό serious infringement γιατί μπορεί να ελεγχθεί αργότερα σε άλλη περίπτωση. Καλύτερα λοιπόν να θεωρήσουμε ότι αν κανείς αρνηθεί τον έλεγχο ακριβώς το ίδιο με τις σοβαρές παραβιάσεις. Να το ξαναδείτε το δεύτερο πίνακα, γιατί είναι ασυνεπής. Ευχαριστώ, Βέρνερ Κούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αλλάζουν οι καιροί, βλέπετε. Πριν από 20 χρόνια οι Ολλανδοί ήταν ε, ηγέτες στην Ευρώπη, ήταν οι πρωτοπόροι. Ναι, ναι, ε, κάπως. Τώρα θέλουν ε, περισσότερες ρυθμίσεις, πιο αυστηρές, όχι μόνο τα τεχνικά, αλλά και τους χρόνους ανάπαυσης και εργασίας. Και τότε στη Γερμανία το συζητούσαμε εμείς στην Επιτροπή Μεταφορών, αν είναι παράτυπο αντί ένα τόνο ε, καύσιμα ε, να έχεις δύο τόνους όπως είχαν οι Ολλανδοί γιατί βάζανε βενζίνη στη Royal Dutch Shell στην Ολλανδία, στο Ρότερνταμ και αλωνίζανε στην Ευρώπη χωρίς να ξαναφουλάρουν. Τώρα λένε «Α, ίσες ε, ευκαιρίες, ίσες δυνατότητες, υποχρεώσεις» και πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Στην Ευρώπη ε, θα πρέπει όλα να γίνονται ομοιόμορφα και ενιαία. Και να μην ε, λέει κάθε υπηρεσία μεταφορών αρμόδια στη Γερμανία ε, ότι εντάξει δεν τρέχει και τίποτα με τους χρόνους ανάπαυσης και μετά η Ολλανδία είναι πιο αυστηρή, η Πολωνοί τελείως διαφορετική. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικός αυτός ο κατάλογος. Ότι έχουμε τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά και για τις κυρώσεις και για τις ποινές και τα πρόστιμα. Και χρόνια οδήγηση και ανάπαυση εκτός από τους τεχνικούς ε, ελέγχους, εκτός από τους ελέγχους του φορτίου και τις άδειε. Ε, ε, είναι σημαντικό, αλλά και τα διπλώματα οδήγηση θα πρέπει να είναι συγκρίσιμα. Αυτό αφορά τις δικές μεταφορές ε, που είναι το α και το ω γιατί είναι ο υπαριθμόν ένα κίνδυνο στους αυτοκινητοδρόμους στα φορτηγά. Αυτά. Κατά τα άλλα, σωστά και χρήσιμα και απαραίτητα αυτά που μας φέρατε, ενα τέτοιο κατάλογος, αν το κοιτάξετε, αν υπερβεί κανείς το δεκάωρο ημερήσιας οδήγησης, ε, τι γίνεται, δεν είναι τόσο δραματικό αν προβλέπετε ε, αλλά αν είναι κατά 15 και πλέον τις 100 είναι σοβαρή παράβαση και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Και υπεύθυνο πάντα είναι ο οδηγό, φυσικά. ποιο θα είναι. Είναι γεγονό αυτό. αυτό οδηγεί. Δεν λέω και η μεταφορική εταιρεία φέρει κάποια ευθύνη, αλλά ο κύριος υπέτειο και ο οποίο θα πρέπει να πληρώσει και να τιμωρηθεί είναι ο οδηγό. ο οποίο συλλαμβάνεται, ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει ε, υφίσταται κάποια κύρωση. Στο καμποτάζ, αν το δούμε έτσι λογικά, σε μια εσωτερική αγορά στην Ευρώπη είναι απολύτως απαραίτητο να συμφωνήσουμε. Γιατί κάνουμε μεγάλες κλιματικές διασκέψεις στο Παρίσι και μετά κυκλοφορούν τα φορτηγά άδεια. Γιατί όχι στο καμποτάζ. Ωραία, πάνε, ξεφορτώνουν και γυρνάνε και να πίσω. Και έχουν χρόνους ανάπαυσης, οδήγησης, μηδενίζουν και το ταχύμετρο και έρχονται, ε, το χιλιομετρητή δηλαδή, και έρχονται και ξαναφορτώνουν. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ανοησίες. Ε, ναι, στην διάνοιξη αγοράς, αλλά κοιτάξουμε και το καμποτάζ. Είμαστε μία Ευρώπη, ένας οικονομικός χώρος. Έχουμε 12,5-3 ΑΕΠ όσο και οι Αμερικανοί και η Νοτιοανατολική Ασία και αν τα καταφέρουμε αυτά θα έχουμε πετύχει πολύ. Ακούω τους συναδέλφους από την Ολλανδία και την Τζάκη που λένε θέλουμε πιο απλές ρυθμίσεις αλλά να ισχύουν για όλους. Αυτά. Ε. Να δούμε και τους longliner που λέει ο Φαντάλιν, αυτά τα γίγας φορτηγά, τεράστια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι όλοι μας ε, συμφωνούμε σε ό,τι αφορά τους ε, κανόνες που αφορούν τους οδηγούς. Όλες αυτές είναι λύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών πέρα από το θέμα του καμποτάζ δεν εφαρμόζονται πάντοτε οι κανόνες με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Διαπιστώνω στη συζήτηση ότι φύγουμε το θέμα του κοινωνικού ντάμπινγκ Υπάρχουν προβληματισμοί για θέματα ανταγωνισμού. Νομίζω ότι εάν έχουμε αυτούς τους προβληματισμούς δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε τίποτα. Το κόστος διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη. Οι αμοιβέ διαφέρουν δεν είναι το ίδιο το κόστος ε, για να γίνει μια μεταφορά στην Ολλανδία ή σε μια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Βεβαίως ε, στην ενιαία αγορά υπάρχει ο ανταγωνισμός που έχει κανόνες, είναι απαραίτητος ο ανταγωνισμός. Στόχος μας είναι να αποφευθεί η δημιουργία κυρίαρχων θέσεων. Πολύ συχνά αναφερόμαστε και στο θέμα των απολαβών σε σχέση με το κοινωνικό ντάμπινγκ. Δημιουργούνται εταιρείε που έχουν την έδρα τους σε μια χώρα, προσλαμβάνουν ε, ε, οδηγούς ε, από μια άλλη χώρα αυτό συμβαίνει και στη Γερμανία και στις κάτω χώρες και με σκοπό τον περιορισμό των, του κόστους. Αυτή είναι μια γνωστή πραγματικότητα σε όλους μας. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε να μας επηρεάσουν πολύ τα προβλήματα του κοινωνικού ντάμπινγκ, γιατί ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί αυτή η πραγματικά ενιαία Ευρώπη που να χαρακτηρίζεται από συνοχή. Ευχαριστώ. Έχω εγγραφεί και εγώ ο τελευταίος κλείνει ο κατάλογος. Γι' αυτό το τελευταίο λοιπόν είχα εντατική συζήτηση με τον Πολωνό Υπουργό Μεταφορών και λέει δεν υπάρχει πρόβλημα αν έχουμε ελεύθερο ανταγωνισμό. Και στη Γερμανία οι Πολωνοί κυκλοφορούν, αλλά τους πληρώνουν με πολωνικούς μισθούς και όχι το μισθό της χώρας. Και ας πούμε λοιπόν ότι αυτό ισχύει και σε τρία χρόνια δεν έχετε πια οδηγούς φορτηγών στην Πολωνία γιατί είναι χαμηλότερη μισθή στη Ρουμανία. Και έρχονται οι Ρουμάνοι και ε, κυριεύουν τη δική σας αγορά. Θα σας άρεσε αυτό, πώς το βλέπετε. Έχω κάποιες αφιβολίες. Γι' αυτά θα πρέπει πάντα να τα έχουμε υπόψη. Και βέβαια θέλουμε να υπάρχουν δυνατότητες διασυνοριακής εργασίας, αλλά του αφορά όλους. Δεν είναι πρόβλημα να το λύσει. Μπορεί να σε βρει και σένα το πρόβλημα. Γι' αυτό υπάρχει στον καποτάζ ε, μια νομοθεσία και κανόνες, αλλά αυτή, η νομοθεσία και οι κανόνες που δεν ελέγχονται, καλύτερα ξεχάστε τους. Γι' αυτό χρειάζεται έλεγχη. Δεύτερο, ποιος είναι υπεύθυνο, ο οδηγός ή η εταιρεία. Πήγαμε ε, σε ένα σταθμό ελέγχου, ε, ένα checkpoint της αστυνομίας και μας είπανε ότι συνέχεια μας τηλεφωνούν, χτες για παράδειγμα, τηλεφώνησε ένας οδηγός, παρακαλώ ελέγξτε με. Γιατί με 17 ώρες στο τιμόνι, το μεροκάματο του τρόμου ε, και ε, μου απαγορεύει το αφεντικό μου να κάνω ε, διάλειμμα, γιατί πρέπει να πάω να ξεφορτώσω. Και βέβαια είναι υπεύθυνο ο οδηγό, αλλά τι να κάνει, άμα πάει και το καταγγείλει και παραπονεθεί στο αφεντικό, την άλλη μέρα θα τον απολύσουνε. Όταν όμως σε μία εταιρεία ε, όλα τώρα τα πρόστιμα 10 με 15% τότε θα πρέπει να ε, πίπτει η ράβδος διότι η παρανομία δεν να επιβαβεύεται, τιμωρείται. Για το δικό πακέτο το συζητάμε μισή ε, μισό χρόνο. Η κυρία Μπόλτς, επίτροπος, πραγματικά ποντάρει στο να έρθει αυτή η πρόταση. Η δέσμη είναι σχεδόν έτοιμη. Αλλά τώρα έχουμε νέα ιεραρχία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουν και πολλά να πούνε οι, ε, επίτροποι δεν έχουν πολύ λόγο, μετά είναι οι αντιπρόεδροι και μετά στην κορυφή είναι Juncker και Τίμερμανς. και αυτοί αποφασίζουν no regulation και better regulation. Και εδώ και μισό χρόνο ή εννιά μήνες τα ξέρω και τα λέω για τη δέσμη του αδικού πακέτου και στον Τίμερμανς και στο Γιούνκερ και μου λένε πάει καλά. Ωραία, άμα πάει καλά έξι μήνες Γι' αυτό, Ισμαήλ, μιλάμε για την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εμπιστοσύνη. Θα απαντήσει η Επιτροπή. Ε, είναι κάτι το οποίο δοκιμάζεται. Μιλάμε για εμπιστοσύνη, αλλά δεν ταυτίζεται αυτή με την προσωπική μας εμπειρία. Λοιπόν, τι κάνετε, έχετε πάρει το OK τώρα το, του κυρίου Σεύκοβιτς ή του κυρίου Τίμερμανς ή του κυρίου Γιούνκερ, ότι θα έρθει αυτή η δέσμη, γιατί να περιμένουμε μέχρι τα τέλη του 2016, αφού είναι όλα έτοιμα σχεδόν. Και όταν είναι έτοιμα και μας λέτε πιθανώς τέλη του έτους, εγώ είμαι 11 χρόνια εδώ, όταν λέμε πιθανώς τέλη ε, του 16, θα χαρώ να έρθει τέλη του 17. Λοιπόν, είτε συμφωνούμε να έρθει τώρα το πακέτο και να κατατεθεί, είτε διαφωνούμε. Αλλά να τα πούμε και ο καθένα να αποφασίζει και να αναλάβει τι ευθύνε του και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τα πείτε και στην ιεραρχία σα εκεί. Και τι θα περιμένουμε άλλα δύο-τρία χρόνια το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε και περιέργεια. Παρακαλώ. Thank you. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι ότι είναι σαφές το μήνυμα που λάβαμε σήμερα. Αυτό το σχέδιο κανονισμού, αυτός ο κατάλογος παραβάσεων είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά μόνο ένα πρώτο βήμα. Εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες έτσι ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με όλους τους κανόνες και όχι μόνο με αυτούς που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια. Αυτός είναι ένας στόχος που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και ο στόχος του θεμητού ανταγωνισμού και η εξασφάλιση δίκαιων συνθήκων εργασία, σωστών συνθήκων ασφαλείας. Συνεπώς, ε, στόχος μας στο μέλλον είναι να εξασφαλίσουμε συμμόρφωση με τους κανόνες, κυρίως αυτούς που αφορούν το καμποτάζ. Θα πρέπει να γίνει και μία αναφορά που αφορούν τα κριτήρια εγκατάσταση και την καταπολέμησης των αποκαλούμενων letterbox companies. Σε ό,τι αφορά την ε, πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε από την Επιτροπή και από τον αρμόδιο Επίτροπο, ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω όπως το έκανε και η Επίτροπος, ότι όλοι κινούμεθα προς αυτή την ανάπτυξη αυτής της πρωτοβουλίας και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι μία εκ των υστέρων αξιολόγηση του υπαρχόντων κανονισμών έτσι ώστε να έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι σαφής, ότι είναι σωστή και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια εξασφάλιση ότι θα μπορέσουν να τεθούν σε εφαρμογή. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο 1071 του 9 και ο 1072 ε, για την πρόσβαση στην ε, αγορά αποτελούν μέρος αυτής της άσκησης της εκτονιστέρων των αξιολόγησης που θα έλεγα ότι έχει προχωρήσει αρκετά και νομίζω ότι με βάση αυτή την αξιολόγηση να ξεκινήσουμε ε, την ε, αξιολόγηση. Δύο παρατηρήσεις που έγιναν εδώ ως προς συγκεκριμένα θέματα που αφορούν το κατάλογο που αναφέρθηκε από τον κύριο Ρίκε σχετικά με τις ενδεχόμενες διαφορές ε, στην σοβαρότητα ορισμένων παραβάσεων, το θέμα των πλαστών των εγγράφων και την παράβαση που αφορά την άρνηση ε, επίδειξης των ε, εγγραφών ιδιαίτερα την παράβαση της ομάδας 2, δηλαδή πλαστά έγγραφα και άρνηση επίδειξης εγγράφων. Θα έλεγα ότι αυτά Τοποθετούν στο ίδιο επίπεδο. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε την άρνηση επίδειξη των εγγράφων ως σοβαρό, σοβαρή παράδοση γιατί οδηγεί στην ε, αλλαγή του παρατήματος 4, κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε δίχως μια πράξη εφαρμογής. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του κυρίου Βαντάλεν σε ό,τι αφορά τα πλαστογραφημένα έγγραφα. Κατά την άποψή μου, τα πλαστογραφημένα έγγραφα όντως αποτελούν μέρος της σειράς παραβάσεων. Θα ήθελα να, να αναφερθώ στον κανονισμό που αφορά την άδεια οδήγησης. Ε, όλες αυτές οι παραβάσεις αναφέρονται τις παραβάσεις της ομάδας 2. Είναι η 8 και η 9. Και αυτό αφορά και τις παραβάσεις της ομάδας 10 και 11 σχετικά με την πλαστογράφηση των εγγράφων. Τελειώνοντας θα μπορούσα να πω ότι το κείμενο αυτό είναι πολύ τεχνικό, πολύ πολύπλοκο και για το λόγο αυτό το ε, ετοιμάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες ένα non-paper, <clears throat> ελπίζω να είναι χρήσιμο. Αυτό προσπαθεί να εξηγήσει τη λογική των παραβάσεων και εξηγήσει μερικές νέες παραβάσεις που ε, συνδιορθώσαμε ή συμπεριλάβαμε σε αυτό τον αναθεωρημένο κατάλογο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω το εξή. Οι ενστάσεις και αντιρρήσεις μπορούν να καταδεθούν μέχρι τις 14 πρώτο 2016 εδώ στη Γραμματεία σε εμάς και στην Ολομέλεια 28 Φεβρουαρίου ψηφίζουμε. Όλα αυτά είναι το αργότερο, είναι η προθεσμία κατάληκτική. Πάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Παρουσίαση από τον κύριο ε, Μίλη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Και θα ήθελα να θυμίσω ότι είχαμε επίσκεψη στη Λισαβόνα, η κυρία Κίλονεν και ο Ρόμπερτ Ζήλε είχαν μεταβίδει εκεί. Έχουμε δηλαδή γνώση για το τι συμβαίνει στον οργανισμό ΕΜΣΑ. Υπάρχει και έκθεση πεπραγμένων. Παρακαλώ, όσοι δεν θέλετε να ακούσετε τη συζήτηση, να αποχωρήσετε. Also, zunächst mal begrüße ich sehr herzlich den... Καλώς ορίζω θερμά τον εκτελεστικό διευθυντή ε, Μίλη, διευθύνοντα σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Οργάσμου για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Οι συνάδελφοι Κίλονεν και Ζήλε ήρθαν, τους γνωρίζετε. Θέλουμε βέβαια και οι υπόλοιποι να μάθουμε τι γίνεται και υπάρχει και μια έκθεση της αποστολής που μοιράσαμε στα μέλη στα πλαίσια του προγράμματος εργασίας του οργανισμού σας. Έχουμε κάποια ενημέρωση ήδη. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε και σας δίνουμε αμέσως το λόγο. Ε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση ξανά εκ νέου σήμερα που μου δίνει την ευκαιρία να σα πω μερικά λόγια για τις δραστηριότητε του ΕΜΣΑ και τις προκλήσεις για το μέλλον. Επαναλαμβάνω ότι είμαι ευγνώμων στην Επιτροπή σας που υποστήριξε τόσο πολύ και βοήθησε τη δουλειά της ΕΜΣΑ από τη δημιουργία της το 2002. Αντίθετα από πέρυσι, φέτος θα ήθελα να τονίσω ποιε είναι οι κύριες προτεραιότητες και προκλήσεις της ΕΜΣΑ στον, για το επόμενο έτος. Αφού μιλάμε λοιπόν για προκλήσεις, η κύρια είναι ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων. Γιατί έχουμε αναγνωριστεί ως κύριο εργαλείο για τη συλλογή γνώσεων και χορήγηση τεχνικής βοήθειας στα κράτη-μέλη, υπηρεσίες της Κομισιόν και άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης. Εδώ βλέπετε ότι η υπηρεσία άρχισε από την αρχή ήδη να εφαρμόζει το στόχο της μείωσης που έθεσαν τα κοινωτικά όργανα και ξεπεράσαμε ακόμα τους στόχους αυτούς. η αριθμοί όμως και το μέγεθος του καθήκοντος αυτού συνεχώς αυξάνονταν. Φτάσαμε τώρα σε ένα σημείο όπου η περαιτέρω μείωση των ανθρωπίνων πόρων θα σήμαινε λιγότερες προτεραιότητες ή περισσότερη στοχοποίησή τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω. Σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στην πρώτη μας μελέτη για τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων και το 16 μας ζητήσατε και θα κάνουμε μια εξωτερική αξιολόγηση όπως προβλέπεται από το καταστατικό μας. Η πολύτιμη συμβολή σας είναι κάτι που το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Στην έμσα η ασφάλεια των πλοίων βρίσκεται στην καρδιά των δραστηριοτήτων μας και αφορά ιδίως την ασφάλεια των επιβατών το 2016 τα αποτελέσματα της μελέτης της ΕΜΣΑ θα γίνουν επί τη βάση πρότασης της Κομισιόν για την ε, περισσότερη ασφάλεια στα πλοία και θα κάνουμε και μια μελέτη για την ασφάλεια κατά των πυρκαϊών για τα επιβατικά πλοία. Θα συνεχίσουμε δε να στηρίζουμε τεχνικώς τη δεύτερη φάση του λεγόμενου fitness check των επιβατικών πλοίων. Όταν κάτι πάει στραβά, και δυστυχώς αυτό συμβαίνει, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΜΣΑ, αυτό γίνεται συχνότερα, όλο και συχνότερα, πέρυσι 3.000 ατυχήματα σημειώθηκαν και δυστυχήματα. 99 σοβαρά, 136 νεκροί και 51 απώλειες πλοίων. Πρέπει από τα λάθη μας να μαθαίνουμε και να προβλέπουμε τέτοια ατυχήματα. Η συλλογή λοιπόν των στοιχείων για τα ατυχήματα και δυστυχήματα αυτά είναι σημαντικό εργαλείο. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε τον κατάλογο των θαλασσίων ατυχημάτων κλπ. Και ο κατάλογος αυτός είναι χρήσιμος και για το κοινό, το βρίσκουμε στην ιστοσελίδα μας. Το 2016 θα συνεχίσουμε να χορηγούμε βοήθεια στα κράτη-μέλη και την Κομισιόν για την εφαρμογή της διεθνούς νομοθεσίας και αυτό θα συμπεριλαμβάνει τη στήριξη, τη βελτίωση για την εφαρμογή των εγκαταστάσεων ελιμενισμού και την ανάπτυξη εναλλακτικών καφουσίμων. Ναι. Υπάρχει και η σχετική οδηγία κανονισμός για το θείο, για τις εκπομπές διοξιδίου και εδώ θα βοηθήσουμε την Κομισιόν και για την ανακύκλωση των πουλίων. Η ΕΜΣΑ είχε εφαρμόσει το σύστημα θέτης, της θέτηδος για όλα αυτά. Η θέτης θα αναπτυχθεί το 16 ως ενωσιακό σύστημα πληροφόρησης για ανταλλαγή πληροφοριών και για καλύτερη στόχευση στο μέλλον των ελέγχων που προβλέπονται ή της συμμόρφωσης με τους κανόνες. Η αναθεωρημένη οδηγία για το θείο ήταν το πρώτο <laughs> καθήκον που αναλάβαμε. Μόλις μέσα σε τρεις μήνες το εφαρμόσαμε αυτό και σε άμεσο μέλλον το θέτης θα γίνει το μοναδικό σύστημα πληροφόρησης για αυτά τα θέματα στην Ένωση και την επαλήθευση της συμμόρφωσης το MRV, ο κανονισμός MRV και ο κανονισμός για την ανακύκλωση των πλοίων είναι τα επόμενα, η επόμενη στόχη μας. Επίσης του χρόνου θα έχουμε νέους εταίρους για να προσεγγίσουν και τρίτες χώρες την νομοθεσία της Ένωσης στην Μεσόγειο, στην Κασπία, στη Μαύρη Θάλασσα θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Το προσωπικό αυτό δεν το εκπαιδεύει μόνο η ΕΜΣΑ, δεν το εκπαιδεύει μόνο η ΕΜΣΑ, αλλά εκπαιδεύει και τα, το προσωπικό των πλοίων που περιμαζεύουν πετρέλαια στη θάλασσα η μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα και των εμπορικών μεταφορών μας απασχολεί επίσης. Το 2016 μετά από διαβούλευση με τις τελωνιακές αρχές ένα πειραματικό πρόγραμμα απλοποίησης και εναρμόνισης των διαδικασιών θα αρχίσει. θέλουμε να αποδείξουμε ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται μπορούν να συμμορφωθούν με το λεγόμενο τα Μανιφέστο». Υπάρχουν και οι νέες τεχνικές επιλογές που έχουμε τώρα και διατίθενται στα ενωσιακά όργανα. Οι προσπάθειές μας έχουν έναν και μόνο στόχο οι κύριοι ενδιαφερόμενοι στον τομέα να έχουν όσα στοιχεία τους είναι απαραίτητα. Η ΕΜΣΑ χορηγεί και υπηρεσίες επιτήρησης στοχευμένες σε συνδυασμό με το Φιρόντεξ για συνεργασία στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Η υπηρεσία λειτουργεί από το 2013 και το Μάιο του 16 θα ανανεωθεί, θα αρχίσει ένα καινούργιο κύκλο. Με στοιχεία για την καλύτερη παρακολούθηση της κυκλοφόρησης των πλοίων. Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν ταχύτερη πληροφόρηση αλλά και άλλα ωφέλη. Και γι' αυτό συμμετέχουμε σε πειραματικά προγράμματα για να δούμε τη δυνατότητα καλύτερου συνδυασμού των εξαποστάσεως ελρομολογίων. Έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την κατάσταση και την κυκλοφορία των μικρών πλοιαρίων που χρησιμοποιούν και οι μετανάστες. Θέλουμε να οθήσουμε αποστολές και επιχειρήσεις με πολλαπλούς στόχους. Επιτήρηση εκπομπών, ε, μόλυνση από έκχυση πετρελαίου κλπ. κλπ. Άλλο σημαντικό σχέδιο από την έμσα του χρόνου θα είναι η εφαρμογή του Κοπερνίκου θα υπογραφεί η συμφωνία αυτή σήμερα και το 16 θα αρχίσει η εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Η υπηρεσία θα πάρει 40 εκατομμύρια κατά την πενταετή περίοδο και η πρώτη φάση τι και θα συνεχίσουμε να επιτηρούμε ενεργά και τη μόλυνση από έξι πετρελαίου στη θάλασσα. Έχουμε 19 σταθμούς επιτήρησης. Από τον καλοκαίρι του 16 θα καλύψουμε και την θαλάσσια περιοχή γύρω από τα Σκαναρίους. Όλα αυτά γίνονται με κοινοπραξία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Εμείς χορηγούμε και τις εγκαταστάσεις για την εποπτεία. Οι ιδιοκτήτες των πλοίων βέβαια έχουν δική τους ιδιωτική εμπορική δραστηριότητα, αλλά έχουν υπογράψει πολλές φορές συμβόλαια με την ΕΜΣΑ. Δηλαδή εθελοντικός θα εγκαταλείπουν την εμπορική τους δραστηριότητα και θα συμμετέχουν σε επιχειρήσεις συλλογής πετρελαίου. Επίσης προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια σειρά υπηρεσιών για τον καλύτερο δυνατό μηχανισμό top-up σε εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου στη θάλασσα όπου μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Για τον μηχανισμό ανταπόκρισης της μολύνσης. Σε αυτή τη φωτογραφία μπορείτε να δείτε το σκάφος της ΕΜΣΑ με δυνατότητα παρέμβασης. Ελπίζω ότι αυτή η αναφορά στις προτεραιότητες και στις προκλήσεις σας έδωσε μία ιδέα του τρόπου λειτουργίας της, ε, ε, του φορέα μας για τους επόμενους μήνες. Ε. Είμαι εδώ για να ακούσω τις ερωτήσεις σας και θα ήθελα να επαναλάβω την πρόσκλησή μου να μας επισκεφτείτε στη Λισαβόνα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much as well. Και, εγώ ευχαριστώ. Μετά από όλη αυτή την ωραία φωτογραφία ε, θα δώσουμε το λόγο όχι με τη σειρά των πολιτικών ομάδων αλλά με τη σειρά φωτογράφησης. <laughs> Το Ρόμπερτ Ζήλε πρώτα. Uh, uh, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν από μερικούς μήνες επισκέφτηκα την ΕΜΣΑ στην ε, Λισαβόνα και πραγματικά με εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Να μην ξεχνάμε ότι ο Μομιντίκα αποτελεί το σύμβολο της ΕΜΣΑ. Θα ήθελα τώρα να περάσω σε κάτι σοβαρότερο. Πραγματικά με εντυπωσίασε ο επαγγελματισμό όλων όσων συμμετείχαν και που μας έδωσαν απάντηση σε πολλά ερωτήματά μας. Ερωτήματα που είχαν ε, σχέση με τη συνεργασία, ΕΜΣΑ, Frontex. Πραγματικά οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν ιδιαίτερα επαγγελματικές. Η δεύτερη εντύπωσή μου είναι ότι γνωρίζετε την χρήση των ε, τεχνολογιών που σας επιτρέπουν να βλέπετε οποιοδήποτε σκάφος, οποιοδήποτε σημείο. Βεβαίως εδώ θα, μιλάς, θα μιλήσουμε και για τα drones, θα μιλήσει η παρακαθήμενη συνάδελφός μου. Η κυρία Φώστερ. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη η εταιρεία σας σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα, ε, ε, δυστυχήματα και τη διερεύνηση των δυστυχισμάτων. Το ερώτημά μου είναι ότι το Δεκέμβριο περιμένουμε ως την Επιτροπή μια τέταρτη οδηγία. Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε τα πράγματα σε ό,τι αφορά αυτή την νομοθεσία. Θεωρείτε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα για τα οποία θα απαιτηθεί και ανθρώπινο και υλικό δυναμικό, εάν δηλαδή η νομοθεσία κινηθεί προς μια διαφορετική κατεύθυνση ε, από ό,τι προτείνει η Επιτροπή. Ξέρετε τη θέση του Κοινοβουλίου, ξέρετε τη θέση του Συμβουλίου. Ε, υπάρχουν ορισμένοι τομείς όπου Ενδεχομένω χρειάζεται νομοθεσία για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων. Ευχαριστώ η Μαρία Κίλωνεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μιλή που ήρθε εδώ και μας ενημέρωσε για την ΕΜΣΑ παρέχοντας καινούργια στοιχεία. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα, πάρα πολύ σημαντικά τα όσα ακούστηκαν και χαίρομαι πάρα πολύ που δόθηκαν πληροφορίες εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι αυτή που αφορά το περιβάλλον και τη θάλασσα. Ξέρουμε για την, τα περιοδηγίες για το θείο, ξέρουμε το θέμα της θαλάσσιας ρήπανσης, πώς φαντάζεστε ότι θα είναι ο, ο ρόλος σας στην θάλασσα, πώς θα μπορούμε να ελέγξουμε το τι κάνουν αυτοί που κινούνται στη θάλασσα και πώς θα μπορούσατε να κάνετε κάτι για τις περιβαλλοντικές αυτές προκλήσεις. Η άλλη μου ερώτηση αφορά τους πρόσφυγες και το κλίμα. Το πρόβλημα που έχουμε τώρα είναι μικρό. Ας σκεφτούμε τι θα γίνει στο μέλλον σε ό,τι αφορά το κλίμα σε μικρές χώρες, σε μικρά νησιά. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα πώς θα μπορούσατε να είστε περισσότερο προετοιμασμένοι για αυτές τις προκλήσεις που διαφαίνονται στον ορίζοντα. Uh, Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Μιλή, ε, για την ε, παρουσία σας εδώ. Έχετε λόγους να είστε ικανοποιημένο χωρίς καμία αμφιβολία για όλα αυτά που έχετε κάνει και για τη ζέση που δείχνετε πάντα στην Επιτροπή μας από τότε που έχει αρχίσει να δουλεύει ο οργανισμός, αλλά είναι και αμοιβαίο. Εμείς ε, συχνά αμφισβητούμε και είμαστε καχύποπτοι απέναντι σε οργανισμούς. Αλλά ε, πάντα ε, η Επιτροπή μας ήταν στο πλευρό σας και έχει επιβεβαιωθεί, έχει δικαιωθεί. Και ήταν, είσαστε πολύ άξιος και στη δουλειά σας. Επανειλημμένα ε, ήμουνα εγώ ε, εισηγητής για δικά σας θέματα. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω στην τελευταία επίσκεψη, αλλά είχα στα εγγένειά σας στη Λισαβόνα. Καθ' όλη λοιπόν τη διάρκεια της ύπαρξής σας, η δική μας Επιτροπή σας ε, υποστήριζε για νέους πόρους και για νέα καθήκοντα. Τώρα, δεν ξέρω είναι καλό ή κακό. Αλλά ακούω από τη μια ότι έχετε βελτιστοποιήσει ε, τους ανθρωπίνους πόρους και έχετε μειώσει το προσωπικό χωρίς να μειώσετε τις δυνατότητες εργασίας σας. Ε, είναι θετικό αυτό, ε, εξακολουθεί να είναι θετικό γιατί κάπως κατάλαβα από όσα μας είπατε ότι έχετε κάποιες αφιβολίες. Αν σας αρκούν οι υπάλληλοι για τα νέα καθήκοντα μπορεί να είναι και περισσότερα αυτά που σας αναθέτουν. Είναι σημαντικό και στην καταπολέμηση της ρήπανσης μου άρεσε πολύ αυτό που άκουσα ότι έχετε προετοιμάσει ένα ε, σκάφος που θα είναι stand-by και θα παραπλέει ε, στις Κανάριες νήσους. Είναι ειδικά σκάφη αυτά και ζητούν ε, μετά τα κράτη, η ΕΜΣΑ κάποια στιγμή να πάνε να απορριπάνουν την περιοχή. Ε, έχετε κάνει κανέναν απολογισμό. Τι γίνεται με αυτά τα πλοία που είναι stand-by και περιμένουν να πάνε να καθαρίσουν όταν έχουμε πετρελαιοκυλίδες. Υπάρχει ε, λόγος να τα έχουμε αυτά κινητοποιημένα γιατί χάνουμε και δύο σπόρους και καράβια που κάθονται εκεί και περιμένουν. Τι γίνεται με τις νέες τεχνολογίες, μιλήσατε για τα drones, ε, πολύ ωραία, αλλά και δορυφόροι υπάρχουν για να δούμε, να εντοπίζουμε πετρελοκυλίδες και να μην ε, ε, υπάρχουν κάποιοι κακοήθεις που ξέρουν ότι ο πληρώνει και προτιμούν να πληρώνουν για να ρηπαίνουν. Ε, να είναι πιο δύσκολο αυτό λόγω των νέων δυνατοτήτων. Τώρα έχουμε αυτό το ατυχές φαινόμενο των προσφύγων για λόγους πείνας, για λόγους πολιτικούς, είναι κατόμφι και στη θάλασσα. Πνίγονται οι άνθρωποι κυρίως στη Μεσόγειο που είναι η θάλασσα όλων μας, αλλά αφορά περισσότερο τις χώρες του Νότου και τη δική μου προκειμένου. Και στην Ιταλία συμβαίνει αυτό. Ε, ε, εκεί σας ζητούν κάθε μέρα περισσότερη βοήθεια για να σταματήσουν ε, τα σκάφη, να σταματήσουν τα τρομερά ναυάγια και συνεργασία με τη Frontex. Εκεί θα μπορούσατε επίσης να μας πείτε δύο λόγια. Τι σας ζητούν, τι μπορείτε να κάνετε και ποιο είναι το αποτέλεσμα τελικά όλων αυτών των δράσεων μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Ειλικρινά ακολουθήστε αυτό το δρόμο, είναι πάρα πολύ καλός, επιτυχής και υποδειγματικός από τη σκοπιά μας θα πρέπει να σας δώσουμε ειλικρινή συγχαρητήρια και συνεχίστε έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Η Λούση Άντερσον. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σε εξ της ομάδας μας. Γιατί ξέρω ότι αντιμετωπίζετε προβλήματα σε δύσκολο δημοσιονομικό κλίμα και εμείς όσο μπορούμε σας βοηθούμε να έχετε τους πόρους που χρειάζεστε. Θα ήθελα να τονίσω τώρα το θέμα της ασφάλειας. Φαίνεται από τους αριθμούς ότι αυξάνονται τα ατυχήματα και δυστυχήματα. Και θα ήθελα να μου σχολιάσετε μερικά από τα σχετικά θέματα, ιδιαίτερα δε για μας τους σοσιαλιστάς ενδιαφέρει το θέμα το, της εκπαίδευσης και των συνθήκων εργασίας καθώς και της εξίσωσης προς τα κάτω γιατί υπάρχει ο φόβος ότι θα μειωθούν οι ασφαλείς μεταφορές στη θάλασσα για μας αυτό είναι προτεραιότητα είχατε μια επιβεβαίωση από τα στοιχεία ότι αυξάνεται η ανασφάλεια. Κύριε Ζήλε, μπορεί να διαφωνείτε μαζί μου, αλλά αυτά εμάς μας ενδιαφέρουν. Αναφέρατε την, τον κανονισμό για τους λιμένας. Είναι ένα σοβαρό ερώτημα αν θα χρειαστούν περισσότεροι πόροι και για τα λιμάνια, διότι ο κανονισμός αυτός δεν ξέρουμε αν θα αναφέρει τα ελάχιστα όρια ασφαλείας. Ξέρω ότι ακόμα γίνονται διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα, αλλά πολλοί λένε ότι πρέπει να καθοριστούν κατώτατα όρια. Για μένα είναι σοβαρό αυτό το θέμα και οι αμφιβολίες που έχω για τον κανονισμό των λιμένων. Συμφωνώ, είναι θέμα πολιτικής επιλογής, αλλά ενδιαφέρονται πολλές χώρες μέλη για αυτό το θέμα. Κατά πόσον έχει νόημα δηλαδή να υπάρξει τώρα αυτός ο κανονισμός. Και παρακαλώ και τους συναδέλφους να το σκεφτούν καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τζάκι Φώστερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Ευχαριστώ πολύ. Όπως και άλλοι συνάδελφοι, και εγώ είμαι νησιώτησα. Είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο γύρω-γύρω θάλασσα και στη μέσα το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πολύ ε, σημαντικά αυτά που κάνετε για τον κλάδο της ναυτιλίας. Εγώ προέρχομαι από την αεροπορία και ιστορικά ήταν πολύ... Ε, διαφανή η προσέγγιση με την οποία αντιμετωπίζουμε τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα, γιατί έτσι βελτιώνεται η ασφάλεια. Τώρα αυτό από πλευρά επιμελητία είναι πιο δύσκολο να το κάνουμε στη θάλασσα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την πίεση και καλό είναι αυτό που είπατε για τους κανονισμούς και να υπάρχει σοβαρή υλοποίηση και εφαρμογή. Γιατί καμιά φορά στον ωκεανό είναι δύσκολο να φτάσει σε βάθος. Στην κυριολεξία όμως αυτή τη φορά. Για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα drones, μόλις έκανα εγώ μια έκθεση ε, πρόσφατα γιατί έχει ευκαιθεί η χρήση του και στο εμπορικό τομέα και στον τομέα της έρευνας και διάσωσης και όλα αυτά. Το Κοινοβούλιο τα παρακολουθεί πάρα πολύ, έχουμε μια πολύ καλή έκθεση και ελπίζω τώρα να δώσουμε και καλή κατεύθυνση στους νομοθέτες. Δεν θέλουμε υπερβολικές ρυθμίσεις για να μην επιβαρύνουμε πάρα πολύ τον κλάδο και να μην μπορούν οι κατασκευαστές να φτιάχνουν αυτά τα αεροσκάφη. Κάπου υπάρχει πρόβλημα και ήθελα να αναφερθώ. Μιλήσατε για την οδηγία για το θείο Εμείς συζητούμε πολύ συχνά με εκπροσώπους της ναυτιλίας και της κρουαζιέρας και τους απασχολούν αυτά τα θέματα και έχει ανακύψει ένα πρόβλημα και θα το θέσω και υπόψη της επόμενης Ολλανδικής Προεδρίας. Ενδιαφέρονται πάρα πολύ σε τέτοια θέματα ναυτιλιακά. Εδώ υπάρχει μια σύγκρουση, γιατί από τη μία έχουμε την οδηγία για το θείο, έχουμε σχετικά ζητήματα με το πώς ε, μπορούν να ε, αγοράσουν ε, διάφορα υλικά και έχουν ένα εξοπλισμό για να καθαρίζουν τις δεξαμενές. Αλλά έχουμε και προβλήματα με κάποια ντόπια λιμάνια όπου ε, υπάρχουν. Όχι, όχι. Έχουν αυτή ε, τη δυνατότητα, αυτό τον εξοπλισμό, αλλά τους λένε δεν ε, ανταποκρίνεστε στην οδηγία για τη βιότητα των υδάτων, για το καθαρό νερό. Γιατί υπάρχει και ε, αντίστοιχος εθνικός κανονισμός. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτό. Υπάρχουν προβλήματα, λοιπόν, και ό,τι μπορείτε να κάνετε θα βοηθούσε. Δεν υπάρχει. Ελπίζω τελικά να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα και θα τα ξαναπούμε. Ο κύριος Φαν Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μιλή που ήρθατε. Χάρηκα πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και μου άρεσε και θα ήθελα να σας συγχαρώ. Έχετε πάρα πολύ ε, μεγάλο και συνολικό πρόγραμμα εργασίας για τις νέες τεχνολογίες, για το, τα drones, δεν θα σας εκπλήξει γιατί είμαι σκιώδης συζητητής ε, της έκθεσης της κυρίας Φώστερ που, που ανέφερε και η ίδια. Λοιπόν, τι χρειάζεστε από τις ε, ε, αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα δηλαδή, για τα drones, για να βοηθηθεί η δουλειά σας για την μετανάστευση και για να ελεγχθεί η ρήπανση τι περιμένετε ε, από τη δική μας Επιτροπή εμπροκειμένου. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Keith Taylor. I found the button. Jolly good. Hello. Uh, thank you very much, Mr. Mary, for uh, your, Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας, κύριε Μίλη. Πρόθεσή μου ήταν να έρθω το καλοκαίρι στη Λισαβόνα αλλά πήγα κάποια προβλήματα με το γόνατό μου και δεν μπόρεσα να πραγματοποιήσω αυτό το ταξίδι. Πριν από μερικά χρόνια το κοινοβούλιο αυτό ψήφισε έτσι ώστε να δοθούν επιπλέον αρμοδιότητες στην ΕΜΣΑ για την πρόληψη της ρήπανσης στη θάλασσα. Εγώ βλέπω ότι η γεωγραφική, τη γεωγραφική σας κάλυψη την ε, αυξήσατε χρησιμοποιώντας ε, τα ιδιωτική ε, χρήσης σκάφη σας. Έχετε κάποιο πρόγραμμα να επεκτείνετε την παροχή υπηρεσιών. Επίσης η άλλη μου ερώτηση είναι κατά πόσον η ΕΜΣΑ έχει τις απαραίτητες, τα προαπαιτούμενα για να μπορεί να παράσχει αυτές τις υπηρεσίες. Η Κλάουδιο Μοντέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίασή σας. Πραγματικά πάρα, ε, πάρα πολύ πλήρης ε, Κάνατε μία αναφορά στην ψηφιοποίηση των λιμένων και αναφερθήκατε και στις νέες τεχνολογίες. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο και με μεγάλη χαρά άκουσα τα όσα είχατε να μας πείτε. Πραγματικά θα ήταν μεγάλη χαρά για μένα να επισκεφτώ την ε, Λισαβόνα και τις εγκαταστάσεις σας. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις. Το πρώτο θέμα αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αναρωτιέμαι αν έχετε προγραμματίσει δραστηριότητες που αποσκοπούν στη βελτίωση της παρεχόμενης κατάρτισης και εκπαίδευσης, τα περισσότερα ατυχήματα ή δυστυχήματα οφείλονται ή αποδίδονται σε ανθρώπινο σφάλμα. Έχετε προγραμματίσει λοιπόν κάποιες δραστηριότητες σε αυτό το δομέα. Επίσης θα ήθελα να γνωρίζω αν έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Υπάρχει και το θέμα της προσφυγικής κρίσης. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι επιπροσθέτως για την συνεργασία με τη Frontex. Κάνετε αναφορά στο γεωγραφικό ο εύρος παρεμβάσεών σας. Θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε λίγο περισσότερο τις ε, περιοχές στις οποίες εργάζεστε στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας με τις χώρες μέλη του αρχιπέλαγος της Μαδέρα. Θα μπορείτε να μου πείτε πώς καλύπτεται αυτή η περιοχή του αρχιπελάγου. Σε ευχαριστώ. Πέτερ Φαντάλεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Άλλο ένα πεδίο που μας λείπει από ε, το πρόγραμμα Juncker και Team Juncker και αυτά είναι τα agencies, οι οργανισμοί. Έχουν ιδρυθεί πάρα πολύ, συσταθεί πάρα οι οργανισμοί και δεν χάλασε και ο κόσμος, ούτε έχει γίνει καλύτερος. Εγώ είμαι υπέρ της ΕΜΖΑ, το λέω ρητά. Πριν από τρία χρόνια, θυμάστε με τον συνάδελφο Ντίρκ και τον συνάδελφο Κουμουτσάκο είχαμε πάει στη Λισαβόνα και είδαμε πραγματικά ποια είναι η προστιθέμενη αξία της ΕΜΣΑ και φάνηκε και από τη σημερινή παρουσίαση. Αυτός ο οργανισμός έχει αποδείξει τη χρησιμότητά του και πραγματικά ε, χαίρομαι που υπάρχει. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Στην ανάλυση ατυχημάτων και δυστυχημάτων. 99 ε, είναι τα πολύ σοβαρά. Και ερωτώ, αυτή την ανάλυση την κάνουμε εδώ και καιρό. Δεν είναι σημερινό, η χτεσινό αυτό το θέμα. Ε, έχουμε ατυχήματα και δυστυχήματα στην αυτιλία. Θα μπορούσατε να μου δώσετε ένα παράδειγμα Συγκεκριμένα λοιπόν η ανάλυση σας που οδήγησε την τελευταία περίοδο. Γιατί το ρωτάω αυτό. Εσείς που κάνετε αυτές τις αναλύσεις, λόγω αυτών των αναλύσεων μειώνετε τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα, δηλαδή πιάνει τόπο η δουλειά σας. Τα αναλύετε, τα μελετάτε, βοηθάει αυτό στη μείωση. Βλέπουμε συγκεκριμένα ότι έχουν μειωθεί τα χύψη δυστυχήματα και ατυχήματα. Αυτό το ερωτώ μεταξύ άλλων, Πρόεδρε, διότι προσωπικά βλέπω να αυξάνονται κάποια είδη ατυχημάτων ναι, ε, ναι, στην ναι. αυσιπλοεία και ε, αυτά είναι ατυχήματα με καλώδια. Ε, έχει να κάνει με την χρήση διαφόρων αληφτικών εργαλείων τα οποία κόβουν καλώδια με διάφορες στράτες και τα λοιπά. και είμαι περίεργος να δω ε, αν το έχετε αναλύσει και το αναγνωρίζετε αυτό. Έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση. για τέτοια συστήματα μέτρησης, καταμέτρησης και ποντισμένα υποβρύχια καλώδια. Ευχαριστώ, Βέρνερ Κούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ ως Γερμανός βουλευτής. Είμαι αρμόδιος για δύο μεγάλα ε, πελάγι θάλασσες που είναι η Βόρεια Θάλασσα και η Βαλτική. Βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία ο οργανισμός σας και η ασφάλεια στην αυσιπλοεία και στη θάλασσα. Και χρειάζεται πρόληψη για την προστασία του περιβάλλοντος. Και τι γίνεται ε, με ε, το έρμα που ε, χύνουν στη θάλασσα και καθαρίζουν τις δεξαμενές τους στα πλοία με βρώμικο νερό. Θυμάμαι από την Τορνιέ το 1987 ήταν η εταιρεία αυτή που έφτιαχνε τις πρώτες πλυντρίδες και υπάρχουν και κομμάντο αβαρίας με ρημουλκά, με ένα σωρό συστήματα ε, όπως στη Γερμανία ε, ε, το έχουν και οι Ολλανδοί και αλλού, ο συντονισμός αυτών των κομμάντων αβαρίας με τις τεχνικές επιδόσεις είναι δικό σας. Δηλαδή όταν γίνει ένα ατύχημα στη θάλασσα, ένα ναυάγιο, είδαμε στο Βισκαϊκό κόλπο πρόσφατα αυτό το πρόβλημα που είχε το, το πετρελαιοφόρο που είπανε να μην πάει σε λιμάνι, να πάει στην ανοιχτή θάλασσα και έγινε χαμός από το πετρέλαιο και την κοιλίδα που πήγε παντού μετά. Πώς συντονίζεται λοιπόν ε, αυτούς τους καταδρομείς της αβαρίας που τρέχουν να σώσουν την κατάσταση μετά από ένα δυστύχημα. Δηλαδή υπάρχει και πρόληψη και όχι μόνο η θεραπεία. τα μη επανδρομένα σκάφη, τα drones, είναι ένα στοιχείο, αλλά υπάρχει και ένα νέο σύστημα που λέγεται Γαλιλαίος για την παρακολούθηση ε, δορυφορική. Ε, κοιτάω ο χάρτη της Βαλτικής και σε πραγματικό χρόνο βλέπετε να αλωνίζουν εκεί ρωσικά δεξαμενόπλια. Ε, και ε, ε, εκεί στο Γιβραλτάρ, στα στενά του Γιβραλτάρ και στα στενά του Βοσπόρου είναι τα πιο ευάλωτα σημεία. Ευχαριστώ πολύ για την δέσμευση και τη στράτευσή σας. Ευχαριστώ. Γράφηκα και εγώ τελευταίως δύο σύντομες ερωτήσεις. Γνωρίζουμε ότι το βαρύ πετρέλαιο, το μαζού του κοινός είναι πάρα πολύ επιβλαβές για το περιβάλλον είναι απόβλητο, ειδικό απόβλητο και τοξικό απόβλητο και θα πρέπει να ε, ε, το διακινούμε με πολύ προσεκτικό τρόπο ε, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Πότε θα απαγορευτεί, από πότε και μετά το μαζότο αυτό. Υπάρχει εναλλακτική λύση, το ντίζελ, καλά, το οποίο δεν είναι και τίποτα φοβερό, αλλά είναι πολύ καλύτερο από το μαζούτ. Αυτό θα ήταν τεράστια πρόοδος. Μπορεί να είναι ένα ζήτημα χρηματικό αυτό γιατί είναι ένα παραπροϊόν της δίλησης του πετρελαίου και κάτι πρέπει να το κάνουμε. Ε, αλλά μήπως να το σκεφτείτε αυτό. Ε, ε Επίση, είχαμε και κάποια ατυχήματα και δυστυχήματα που αναφέρατε ε, στο Northern Atlantic και στο το Φλαμίνια. Αυτό το ναυάγιο το συζητήσαμε πάρα πολύ εδώ, γιατί δεν ε, ήθελε να βοηθήσει το πιο κοντινό ε, λιμάνι και το γυρίσανε πίσω και ήταν πολύ περισσότερα τα χιλιόμετρα. Εμεί είμαστε ευρωπαϊκό χώρο. Η αμοιβαία συνδρομή και η αλληλεγγύη και η βοήθεια θα πρέπει να είναι ύψιστη προτεραιότητα. Θα τρέξει αμέσω να βοηθήσει. Τι είναι αυτά. Υπάρχουν ε, συνέπειε, Εγώ είμαι δάσκαλο στο επάγγελμα. Αλλά ε, ε, ε συνήθω λέμε ότι μαθαίνουμε αυτά τα σφάλματα μα. Εσεί μάθατε τίποτα από το ατύχημα αυτό Φλαμίνια. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τους ε, βουλευτές που υπέβαλαν τις ερωτήσεις τους. Ο χρόνος πιέζει, θα κάνω μία προσπάθεια να απαντήσω στον εκτενή αυτό κατάλογο ερωτήσεων. Βεβαίως, εάν δεν απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις, μπορώ βεβαίως ε, να αποστείλω ένα email. Θα ήθελα καταρχάς να πω δύο λόγια σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό. Όταν αυτό το ανακοινωθέν της Επιτροπής ε, υπευλήθη το 2013, αρχίσαμε να κάνουμε αυτές τις μειώσεις, γιατί είχαμε απόλυτη συνείδηση ότι όσο πιο νωρίς ξεκινούσαμε, τόσο πιο γρήγορα θα καταφέραμε να κάνουμε αυτή την περικοπή του προσωπικού κατά 5%. Και έχουμε την απαιτούμενη εμπειρία έτσι ώστε να μπορούμε να προσλαμβάνουμε εκτός της εταιρεία. Υπάρχει, έχουμε το απαραίτητο προσωπικό για να ε, μπορούμε να διατηρούμε αυτό το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να καταρτήσουμε το προσωπικό μας, αναδιοργανωθήκαμε, έτσι ώστε να είμαστε στο ύψος των, απε... των προαπαιτούμενων, των απαιτήσεων. Θα πρέπει να πω ότι όλοι οι οργανισμοί διαμαρτύρονται για αυτό το επιπρόσθετο 5% και θα πρέπει μέχρι το 18 να γίνει μια περαιτέρω περικοπή κατά 5%. Συνεχθήκαμε στο Δουβλίνο πριν από ένα μήνα και συζητήσαμε αυτό το θέμα και ενημερωθήκαμε ε, ότι ενδεχομένω αυτό θα μπορούσε να μετατεθεί στο 2020 αλλά είναι προς επιβεβαίωση. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η επιπρόσθετη περικοπή. Δηλαδή ε, θα πρέπει να μειωθεί ο ρυθμός των εργαζόμενων και αυτό είναι πραγματικά μία πρόκληση για μας. Μιλάμε για επτά εργαζόμενους Βεβαίως ε, γνωρίζουμε ποιες είναι οι ανάγκες και ενημερωνόμαστε από τις διάφορες γενικές διευθύνσεις και κατα, καταβάλουμε μία προσπάθεια να λάβουμε υπόψη μας τα όσα μας λένε ε, από τη Γενική Διεύθυνση Περιφάλλοντος, να γίνονται έλεγχοι, να γίνεται ανακύκλωση κτλ. Αυτό σημαίνει μια μεγάλη πρόκληση για τον οργανισμό μας. Βεβαίως μας λείπει το προσωπικό σε ό,τι αφορά τις ε, θέματα σχετικά με τις ε, ενιαίες θηρίδες. Δεν ε, έχουμε την απαιτούμενη πείρα για τα drones. Θα δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα της πρότασης της Επιτροπής. Αν δηλαδή θα υπάρξουν οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι για την ανάπτυξη των drones Ύστερα η διερεύνηση δυστυχημάτων. Αρχίσαμε να, συγκεντρώνουμε, να δημιουργούμε αυτή την βάση δεδομένων που είναι κάτι παρεμφερές ε, με την βάση δεδομένων των αεροπορικών δυστυχημάτων. Έχουμε ξεκινήσει μία ε, πιο προσεκτική ανάλυση των ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Το σημαντικό είναι το να μπορούμε τα δυστυχήματα αυτά να τα αναλύουμε και να αντιδρούμε ε, με τον κατάλληλο τρόπο. Το θέμα όμως είναι η αντίδραση είναι εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων. Αυτές είναι οι βασικές προκλήσεις με τις οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωποι σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Περνάμε τώρα στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Συνεργαζόμαστε με την αρμόδια γενική διεύθυνση, η οποία είναι ιδιαίτερα ευτυχής με την συνεργασία μαζί μας ε, Έχουμε δημιουργήσει το πρόγραμμα θέτης που αφορά τον έλεγχο του θείου και εξελίσσουμε ε, αυτό το μέσο ε, κάνουμε καταλόγους των εκθέσεων ε, που ανεβαίνουν στο σύστημα. Έχουν διεξαχθεί 6.000 έλεγχοι στις χώρες μέλη και θα πρέπει να σας ομολογήσω ότι κατεγράφησαν πάρα πολύ λίγες παραβάσεις σε ό,τι αφορά το θέμα του θείου. Το 2, 2% είναι οι παραβάσεις και οι περισσότερες από αυτές είναι διοικητικού χαρακτήρα. Δηλαδή δεν μιλάμε για παραβάσεις που αφορούν τα καύσιμα. Αφορούν μία μη συμμόρφωση ως προς τις διοικητικές διαδικασίες. Αυτό το κάνουμε κάθε φορά για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Βεβαίως ε, εκπαιδεύουμε τις, ε, τους εργαζόμενους, ε, εκπαιδεύουμε τους άμεσα εμπλεκόμενους σε αυτά τα θέματα. Έχουμε επίσης στενή συνεργασία με την ΕΞΑ και σε τακτική βάση ανταλλάσσουμε πληροφορίες ΕΞΑ και ΕΜΣΑ. Αν κοιτάξετε το θέμα των προσφύγων, θα δείτε ότι είναι ένα θέμα που βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στη μερισία διάταξη και της Επιτροπής. Φέτος πέρασα πάνω από 800.000 άτομα. Συνεργαστήκαμε με την Frontex από το 2013 και τους ε, δώσαμε πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των θαλασσίων συνόρων. Τώρα υποβάλαμε μία πρόταση σχετικά με το πώς μπορεί να αυξηθεί αυτή η δυνατότητα ελέγχου. Μπορούμε να αναπτύξουμε ε, μη επανδρομένα ε, σκάφη και μπορούμε να ελέγξουμε όλες τις πληροφορίες δια δορυφόρου. Εξακολουθούν όμως να παραμένουν μαύρες τρύπες οι οποίες δεν καλύπτονται. Ας πούμε δεν έχουμε δορυφορικές ε, εικόνες, έχουμε ε, χερσαία ή αλλά δεν, δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό. Η χρήση των drones θα μπορούσε να συμπληρώσει τη συγκέντρωση πληροφοριών που θα μπορούσαμε να δώσουμε και στην Frontex καθώς και στις ε, ε, αρχές των χωρών μελών. Τώρα, Σε ό,τι αφορά τα σκάφη ανάκλησης, μιλάμε για 19 σκάφη. Μόλις τελείωσε ο διαγωνισμός, η προκήρυξη στις Καναρίους νήσους και στην Μαδέρα. Αυτό θα, υποφάσισε να εφαρμοστούν το 2016. Με αυτούς τους οικονομικούς πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας κινούμεθα γύρω στις 160 εκατομμύρια για ένα χρονικό διάστημα 7 ετών. Αλλά δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο για άλλα σκάφη. Τώρα βρισκόμαστε σε μια οριακή κατάσταση γιατί θα πρέπει να μας απασχολήσουν και οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου. Έχουμε διοχετεύσει κονδύλια για την παροχή ασφάλειας σε περίπτωση ενός ατυχήματος που ελπίζουμε να μην συμβεί. Έχουμε 8.000 τέτοιες Έχουμε χίλιες τέτοιες εγκαταστάσεις. Έχουμε, έχουμε ένα στο Έχουμε ένα στόκ πάλι στην Πορτογαλία, στην Κύπρο. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ότι έχουμε stockpiles που μπορούμε και στη Μάλτα και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε περίπτωση ατυχήματος. Βεβαίως και η βιομηχανία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα αεροπλάνο. Υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι πάροχοι υπηρεσιών Έχουμε 6 εκατομμύρια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για αυτή τη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια όλου του χρονικού δημαστήματος. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πάρα πολύ περιορισμένα κονδύλια σε περίπτωση ατυχήματος ενδεχομένως ε, θα θυμάστε ε, το μεγάλο ρωσικό αλλιευτικό σκάφος που ε, πήρε φωτιά το κόστος της αντιμετώπισης αυτού ήταν 40 εκατομμύρια. Γι' αυτό και μόνο το λιευτικό σκάφος. Και ήταν ε, ένα περιορισμένο ε, δυστύχημα, σε μεγαλύτερο δυστύχημα. Καταλαβαίνετε ότι ε, τα χρήματα που θα απαιτηθούν είναι πολύ περισσότερα, ας πούμε, αν συμβεί κάτι παρόμοιο με αυτό που συνέβη στο Μεξικό. Τώρα, κατάρτιση. Παρέχουμε κατάρτιση όχι στους εργαζόμενους στον αλλιευτικό κλάδο, αλλά σε προσωπικό από τρίτες χώρες. Υπάρχουν δύο προγράμματα, ένα με τις ε, ε χώρες και ένα άλλο στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Τα προγράμματα αυτά περατώνται του χρόνου, αλλά θα συνεχιστεί αυτή η κατάρτιση σε συμφωνία με τις αρχές. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε να μπορέσουν να, να κάνουν κάτι για την προστασία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει σχέση και με τις, ε, με τις χώρες της και με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε λοιπόν και αυτές οι χώρες να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με μας. Ο χρόνος πιέζει, αλλά να δούμε τι έχουμε κάνει με τους πρόσφυγες. Αυτή είναι μια μεγάλη ε, πρόκληση. Για θυμηθείτε το δυστύχημα Φλαμίνια και την ατυχή κατάληξη από τότε που συμβιώθηκε το δυστύχημα είχαμε μέσα σε σενή συνεργασία με τις χώρες μέλη και με τις επιδεσίες της Επιτροπής και καταβάλαμε μία προσπάθεια να επαναλάβουμε τις κατευθυντήριες γραμμές μας στις χώρες μέλη για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση τέτοιου ατυχήματος. τα κονδύλια μας καλύπτουν λοιπόν το 2016, θα πρέπει όμως να δούμε αν υπάρχει ανάγκη επανεξέτασης αυτής της οδηγίας. Βεβαίως τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν περισσότερο ακριβείς κατευθυντήριες γραμμές από τις χώρες μέλη. Κάποιος έθεσε το θέμα του δυναμικού ελέγχου. Όλα, όλα τα εμπορικά ε, σκάφη τα οποία κινούνται στα θαλάσσια περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχονται από την ΕΜΣΑ. Βρίσκονται στην οθόνη μας οποιαδήποτε στιγμή, ξέρουμε, ξέρουμε από πού έρχονται, εν μέρη ξέρουμε τι εμπόρευμα μεταφέρουν, ε, πού πηγαίνουν κτλ. Και όλο και περισσότερο παίρνουμε πληροφορίες σε γενικότερο επίπεδο, γιατί υπάρχει ο, ο δορυφόρος ΕΕΑΕΣ που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ε, έναν ε, παγκόσμιο, έναν έργο σε παγκόσμιο επίπεδο. Και όταν συνεργαζόμαστε, για παράδειγμα, στην περιοχή του κέρατος ε, της Αφρικής στα πλαίσια του προγράμματος Αταλάντα, προσπαθούμε να χτυπήσουμε την πειρατεία. Έγιναν ορισμένες συζητήσεις στο κόλπο της Γουινέας, αλλά δεν μας ζητήθηκαν, δεν να δώσουμε αυτές τις πληροφορίες. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για τα βαρέα καύσιμα. Εγώ βεβαίως δεν είμαι μάντης, πιστεύω όμως ότι στο μέλλον, ή μάλλον αν κοιτάξετε την καθημερινή ειδησιογραφία, η ναυσιπλοεία κινείται όλο και περισσότερο σε πιο καθαρά καύσιμα στο το ή στη χρήση βιοκαυσίμων χρησιμοποιούν ε, το μεθάνιο. Ναι. Θα πρέπει βεβαίως να γίνουν ε, ε, σεβαστά τα πετούμενα όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά γενικότερα. Βλέπετε ότι υπάρχει μια φθήνουσα χρήση των βαρέων καυσίμων και μέχρι το 2025 πιστεύω ότι θα χρησιμοποιούνται πολύ λιγότερες ποσότητες ε, βαρέων καυσίμων. Αυτό το έχω ξανακούσει πριν από 10 χρόνια το μέλλον. Ναι, αλλά τώρα αυτό ε, όσο περνάει ο καιρός επαληθεύεται. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Κούν, χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο, το 2020 είπαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μουλή που μας ήρθατε και απαντήσατε ερωτήσεις. Ε, would please... Παρακαλώ να σταματήσετε τις ιδιωτικές συζητήσεις ή να φύγετε από εδώ μέσα, ησύχως, να διαλυθείτε. Ορίστε μας. Πάμε στο επόμενο θέμα στη μέση διάταξη. Το οποίο είναι... Δικαιομάδα Δική ομάδα τουρισμού που ανήκει σε αντικείμενο της Επιτροπής μας παρουσίασε από το Γενικό Γραμματέα ε, του ε, Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού του ΟΗΕ. Είναι ο κύριος Ταλέ Μπριφάη. Καλώς ορίσατε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας υποδεχόμαστε. Προηγουμένως θα ήθελα όμως να καλωσορίσω μια ομάδα επισκεπτό του κυρίου Ντουέι που παρευρίσκεται σήμερα εδώ. Καλώς ορίσατε είναι δημοσιογράφη από την Ουγγαρία. <laughs> Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Ταλεμπριφάη, Γενικό Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Δεν είστε εδώ για, για πρώτη φορά βέβαια στην Επιτροπή μας επίσημα, έχουμε ξανασυναντηθεί. Εδώ και καιρό συζητούσαμε τη δική σας επίσκεψη και τώρα χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους τα καταφέρατε και ήρθατε στην Επιτροπή μας. Η συζήτησή μας γίνεται στα πλαίσια της ειδική ομάδας τουρισμού που ήδη από την περασμένη θητεία εσείς η Επιτροπή μας που είναι αρμόδια και για τον τουρισμό. Εκεί συμμετέχουν ε, όλες οι πολιτικές ομάδες με μέλη ε, που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για θέματα τουρισμού. Η ομάδα αυτή ειδική εγκρίθηκε για να υλοποιηθεί η στρατηγική για τον τουρισμό ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να έχουμε μια κοινοβουλευτική παρακολούθηση και έλεγχο, γιατί είμαστε Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού εμείς. Επανειλημμένα το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει ψηφίσματα με τελευταίο εκείνο της έκθεσης συναδέλφου Ντεμόντε που ασχολείται με τις σημερινές προκλήσεις της βιομηχανίας και του κλάδου του τουρισμού στην Ευρώπη. Μεταξύ αυτών γίνεται λόγος και μεταξύ άλλων στην ενίσχυση του τουρισμού στην Ευρώπη, τη διατήρηση της σημασίας και την προώθηση. Όπως ίσως να γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δικαίωμα και εξουσίες εναρμόνισης στον τουρισμό. Αυτό είναι μάλλον υπόθεση των κρατών μελών. Γι' αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό τα κράτη-μέλη στην προώθηση να έχουν ενιαία γραμμή και να κοιτάει ο πέρα από την εθνική του μύτη, που πράγμα δύσκολο ενίοτε. Άρα σημαίνει ενιαία προώθηση του τουρισμού και διαφήμιση στις τρίτες χώρες, ε, προϊόντα καινούρια, διασυνοριακά ή πανευρωπαϊκά για να προσφέρονται σε άλλες περιφέρειες του κόσμου. Τα τελευταία χρόνια η αγορά του τουρισμού έχει γνωρίσει μια μικρή επανάσταση με την ψηφιακή τεχνολογία ε, που επηρεάζει την αγορά και τις συμπεριφορές. Βλέπουμε να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια νέες εταιρείες και ε, παραγωνίζουν παλαιές δομές. Ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις βλέπουν εδώ νέες ευκαιρίες αλλά και αυξανόμενο ανταγωνισμό. Η αηφορία, η βιωσιμότητα, η προσβασιμότητα για όλους, η προσφορά και η ζήτηση είναι θέματα που απασχολούν περισσότερο τον τουρισμό και στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίω. Αυτή ήταν μια μικρή εισαγωγή από πλευρά μα και τώρα με ιδιαίτερη χαρά περιμένουμε να ακούσουμε τα δικά σα. Έχετε το λόγο. Thank you Σας κατευχαριστώ κύριε Κράμερ. Είναι πάντοτε μεγάλη ειδονή να σας συναντώ. Θα αρχίσω λέγοντας πόσο χαίρομαι που έχω αυτή τη δυνατότητα να σας μιλήσω σήμερα. Γιατί ξέρω πολλά πρόσωπα, έχω πολλούς φίλους εδώ μέσα στο κοινό. Και κάθε φορά χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Όνλη. Πάντοτε ζητώ Συγγνώμη αν δεν προφέρω σωστά τα ονόματα, γι' αυτό συγγνώμη κύριε Στεμπάν για τη διοργάνωση της συνάντησης. Επίσης την κυρία Κλαβδία Ντεπαρντέλ. Την συνάντη γνώρισα το πρωί μόλις. Αγαπητοί φίλοι και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του οργανισμού τουρισμού που τους βλέπω ορισμένου εκεί στις πίσω θέσεις. κανά ότι είναι μεγάλη χαρά η συνάντησή μας Η οργάνωσή μας είναι περήφανη για τις καλές σχέσεις που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η σημερινή συνάντηση είναι καμπή. Θα αρχίσω κάνοντας το ιστορικό γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα έχουμε και ερωταπαντήσεις. Αν κάποιος από εσά κοιμήθηκε αργά και είδε τα νέα από την Καλιφόρνια, θα είδε ότι κάθε μέρα ακούμε ειδήσει που μας καταθλίβουν, μας μειώνουν τις ελπίδες, μας απελπίζουν. Αυτό ελπίζω να δείξω με την παρουσίασή μου ότι μπορεί να ανατραπεί. Είναι πλέον καιρός όλοι μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλοι, να συνεργαστούν αν θέλουμε το μέλλον των κοινωνιών μας να είναι ελπιδοφόρο. Ο ΙΕ βασίζεται σε τρεις πυλώνες, κοινωνική πρόοδο, συμπερίληψη, ειρήνη και ανθρώπινα δικαιώματα. Τέσσερις θυλώνες δηλαδή. Που είναι και είναι αρχές και της Ένωσης. Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις παντού μας δείχνουν ότι η τρομοκρατία είναι σφαιρική απειλή και μόνο με συντονισμένη ανταπόκριση μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυνάμεις, τους σκότους, τις σκοτεινές δυνάμεις μεμονωμένα. Ούτε η Γαλλία, ούτε η Ρωσία, ούτε η Τουρκία, ούτε η Τινησία, ούτε η Ταϊλάνδη, ούτε κανένα, καμία άλλη χώρα μόνη της. Είναι επίθεση σε όλους μας. Είναι λοιπόν σφαιρική πρόκληση και χρειάζεται σφαιρική ανταπόκριση. Και αυτό πρέπει να το μεταφράσουμε σε πράξη, σε δράση όταν προσβάλλεται κάποια χώρα, κάποιος προορισμός, πρέπει όλοι μαζί να τη βοηθήσουμε και όχι να την τιμωρήσουμε στοχοποιώντας την. 2. Η κρίση των προσφύγων. Και σε αυτήν μόνο όλοι μαζί μπορούμε να βρούμε μια λύση. Εσείς στην Ευρώπη ξυπνήσατε έγκαιρα και συνειδητοποιήσατε το πρόβλημα. Ταυτίσατε σωστά ότι ποτέ δεν θα μπορέσει να λυθεί αυτό το πρόβλημα μεμονωμένα. Πρέπει να συνεργαστούμε, να εναρμονίσουμε την πολιτική μας, τη στάση μας και να επιμείνουμε στις αρχές μας. Πολύ σημαντικό θέμα που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τρίτον, τη στιγμή που μιλάω συναντώνται φίλοι μας και συνάδελφοί μας στο Παρίσι για το COP21 για την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Ελπίζουμε να καταλήξει σε ιστορική συμφωνία και θα καταλήξει εκεί μόνο αν είμαστε ενωμένοι. Όλα αυτά σημαίνουν ότι χρειάζεται συνεργασία. Δεν μπορούμε τέτοιου είδους προβλήματα που μας δοκιμάζουν να μας διαιρέσουν. Τέταρτον, οι επιπτώσεις της τεχνολογίας έχουν γίνει τόσο σημαντικές ώστε όπως είπε και ο πρόεδρος είναι κάτι αναπόφευκτο να συζητηθεί. Άλλαξαν οι κανόνες του παιχνιδιού. Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε τι ηγετικό ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρώπη εδώ. Οι καταναλωτικές τάσεις επίσης αλλάζουν και οι δυνατότητες μας επικοινωνίας καθημερινά και κάθε λεπτό σχεδόν τουλάχιστον για όσους εξαρτώνται από τα κινητά τους τηλέφωνα είναι κάτι που δείχνει ότι η πληροφόρηση μπορεί να γίνει πολύ γρηγορότερη. Και πέμπτον, οι οικονομικές προκλήσεις δεν έχουν ακόμα λυθεί. Βλέπουμε μια σχετική αναθέρμανση αλλά χωρίς ε, απασχόληση. Χρειάζεται λοιπόν συλλογική δράση για την εκμετάλλευση των νέων τάσεων ή ευκαιριών, ιδίως για τις γυναίκες και τους νέους που δεν βλέπουν κανένα φωτεινό μέλλον μπροστά τους. Πρέπει να ενωθούμε λοιπόν και γι' αυτό. Και γιατί είναι σημαντικά αυτά τα θέματα σε ένα τέτοιο βήμα και σε έναν τέτοιο χώρο. Διότι, τολμώ να πω, το είπα και σε καλή φίλος μου εχθές, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μάλλον μία, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της παγκόσμιας και πανανθρώπινης ιστορίας. Μπορεί να μην το βλέπετε τώρα γιατί είστε μέσα στην ιστορία, αλλά εμείς απ' έξω τη θεωρούμε πολύ ελπιδοφόρο πρότυπο για, τον για ολόκληρο τον κόσμο. Πριν από μερικά χρόνια η Ευρωζώνη αντιμετώπιζε προβλήματα. Σήμερα τα αντιμετωπίζει η ζώνη του Σέγγεν. Πρέπει να τα αντιμετωπίσετε όλα αυτά προς όφελος του κόσμου ολόκληρου. Γι' αυτό η παρουσία μου εδώ και η συνομιλία μας είναι απολύτως σημαντική. Μην τα παρατήσετε, μην μας απογοητεύσετε. Οι προκλήσει μπροστά μας είναι πολλές και περισσότερο από ποτέ χρειάζεται ένωση, ενότητα. Υπάρχουν πάντως και λόγοι αισιοδοξία. Τολμώ να πω επίσης ότι ο κόσμος είναι καλύτερος από ποτέ. Δέστε πόση πρόοδος έχει επιτευχθεί τα τελευταία 40-50 χρόνια από το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου. Θέλω να είστε αισιόδοξοι και να συνδέσω την αισιοδοξία αυτή με την τουριστική βιομηχανία την οποία υπερηφάνως αντιπροσωπεύω εδώ. Παρά την οικονομική ύφεση και τις γεωπολιτικές εντάσεις τα προβλήματα ασφαλείας, ιατρικές κρίσεις, ο τουρισμός ως βιομηχανία συνεχίζει να αναπτύσσεται. Πάνω από οποιαδήποτε άλλη, για έξι συνεχή έτη, η αύξησή του είναι 4,5 με 5% παγκοσμίω, διότι ο τουρισμός δεν είναι απλώς ένας οικονομικός τομέας, είναι πια τμήμα του πολιτισμού και του τρόπου ζωής μας. Και θα συνεχίσει έτσι τον περασμένο χρόνο αυξήθηκαν τα κέρδη από τον τουρισμό κατά πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Σαν να πήγαινε ο καθένας δυο φορές εκτός της χώρας του και να επέστρεφε. Και συνεχίζεται η αυξητική αυτή τάση. Αυτό μας χαροποιεί διότι ενισχύονται έτσι και οι θέσεις απασχόλησης και οι εξαγωγές. Ιδίως σε μια Ήπειρο που θέλει να γίνει σαν την Ευρώπη ηγέτης παγκοσμίω. Πέρα από τα δεδομένα όμως τα στατιστικά στοιχεία, οι επιπτώσεις του τουρισμού είναι και άλλες. Είναι το θεμέλιο της ειρήνης και η καταστροφή των κοινοτοπιών και στερεοτύπων. Αν έχει επισκεφθεί κάποιος κάποιον λαό δεν μπορεί να έχει προκαταλήψεις εναντίον του. Όλα αλλάζουν με τα ταξίδια. Εγώ είμαι καλύτερο άνθρωπος διότι ταξιδεύω και όλοι μπορούν να το έχουν αυτό. Ανοίγει το μυαλό και η καρδιά. Έτσι το βλέπουμε εμείς. Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός προϋπολογισμός του κόσμου. 580 εκατομμύρια την επισκέφθηκαν φέτος είναι και οι περισσότεροι τουρίστες Ευρωπαίοι παγκοσμίω. Αύξηση 5% τους πρώτους 9 μήνες του 2015. Είναι βέβαια νωρίς για να κάνουμε την πλήρη αξιολόγηση των τελευταίων ε, επιθέσεων στον τουρισμό, αλλά η εμπειρία δείχνει ότι τέτοιες επιθέσεις συνήθως δεν έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Και νομίζουμε ότι δεν θα πλήξουν τον τουρισμό της Ευρώπης. Ελάχιστες φορές έπεσε ο τουρισμός. Το 2001 μετά την επίθεση της 11 Σεπτεμβρίου, το 2003 τους επιθέσεις στην Ανατολική Ασία και το 2009 με την χειρότερη οικονομική κρίση που γνωρίσαμε ποτέ. Αυτή τη στιγμή βέβαια προτεραιότητα πρέπει να είναι για όλους μας η ασφάλεια και να θεωρηθεί ως κάτι που δεν μπορούμε να αποφύγουμε αλλά δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται σαν δικαιολογία για να αποκλειστεί ή να μειωθεί ο τουρισμός ή να μας εκφοβήσει για να χάσουμε τη μάχη με τις σκοτεινές δυνάμεις. Ο η χειρότερη ανταπόκριση θα ήταν να σταματήσουμε να ταξιδεύουμε. Ο τουρισμός ε, δείχνει την ε, ομορφιά της διαφορετικότητάς μας. Θα πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Αγαπητοί φίλοι, η Ευρώπη θα πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο σε τρεις ε, τομείς. Η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο γιατί η Ευρώπη χάνει το μερίδιο της αγοράς από τον αναφιόμενο κόσμο. Σε επίπεδο αριθμών η Ευρώπη θα λάβει μόνο το 40% των ε, ταξιδιωτών. Αλλά αυτό δεν είναι απώλεια, γιατί αριθμητικά πάντα μεγαλώνουν και ο, ε, και ο κόσμος ε, γίνεται, θα αρχίσει να ευημερεί όλο και περισσότερο. Μία στις 10 ε, εργασίες αφορούν το τουρισμό, το 9% του ΕΕΠ από το τουρισμό, το 30% του εμπορίου και του τουρισμού, το υπηρεσιών είναι από το τομέα του τουρισμού. Είναι μια σημαντική βιομηχανία και θα πρέπει να μοιραστούμε τα ωφέλη. Η Ευρώπη θα παίξει, πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο πρώτον στον τομέα των κλιματικών αλλαγών. Ξέρω πόσο προσφυλέ είναι για εσά αυτό κύριε Πρόεδρε και αυτό είναι κάτι που το σέβομαι. Οι κλιματικές αλλαγέ βρίσκονται στο επίκεντρο της δέσμευσής μας. Η βιομηχανία του τουρισμού αποτελεί συμβάλλει κατά 5%, όχι 20, όχι 30% στην, ε, στο διοξίδιο του άνθρακα. Θα πρέπει ως τουριστική βιομηχανία να δείξουμε ότι μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτή την τάση. Συνεργαζόμαστε σε πολλά κοινά προγράμματα. Ε, ε ενεργειακά προγράμματα για παράδειγμα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να θέσουμε το σωστό παράδειγμα, να μην θεωρήσουμε ότι η ανάπτυξη είναι ο εχθρός. Ο εχθρό είναι η ανεύθυνη, η μη βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί η ανάπτυξη αυτή δεν δημιουργεί σε δημιουργία εισοδήματος. Η ανάπτυξη δεν είναι ο εχθρός. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλω να τονίσω, γιατί υπάρχουν εκείνοι που μας λένε ταξιδέψτε λιγότερο, κινητοποιηθείτε λιγότερο. Όχι, Μπορεί να υπάρχει βιωσιμότητα από τη μία πλευρά και ανάπτυξη από την άλλη. Μπορούν να υπάρξουν και τα δύο με έναν υπεύθυνο τρόπο. Δεύτερον, η Ευρώπη θα πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο σε επίπεδο επιχειρηματικό. Σήμερα η τεχνολογία άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού. Η, η, η αποκαλούμενη sharing economy ε, αποτέλεσε τη βάση της οικονομίας μας. Ε, σε πόλεις όπως η Βαρκελόνη, το 2 ε, της, ε, ε, των καταλήμματων ανήκουν στην shared economy. Εμείς ζητάμε από την Ευρώπη να παίξει ηγετικό ρόλο. Ξέρω ότι το, ε, η ρύθμιση δεν μας βρίσκει όλους σύμφωνους, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μία οργάνωση. Είναι σημαντικό να υπάρξει μία κοινή βάση. Θα πρέπει να υπάρχει, ε, να συνυπολογίζονται παράγοντες όπως η ασφάλεια, όπως η... Ε, οι άνθρωποι τώρα μοιράζονται τα πάντα, τα σπίτια τους, ε, τα ποδήλατά τους. Ε, υπάρχει δυνατότητα ακόμα και να ε, ε, πα, σε ένα σπίτι και ε, να φας εκεί, να σου προσφέρουν ένα γεύμα. Αυτά είναι νέα φαινόμενα. Δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε. Θα πρέπει όμως να γίνουν με έναν οργανωμένο τρόπο. Τέλος, η Ευρώπη θα πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση του ταξιδιού. Ορισμένοι θα βρουν ε, ότι θα πρέπει να λέμε ότι δεν θα πρέπει να κλείνουν τα σύνορα. Η ασφάλεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Θα πρέπει τα ταξίδια να είναι και φιλικά και ασφαλή. Δεν μπορούμε να θυσιάσουμε το ένα εις βάρος του άλλου. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνουμε. Δεν είναι η στιγμή τώρα για να κάνουμε ότι δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά τα θέματα. Δεν μπορούμε να βλέπουμε χώρες να δαπανούν τόσα ε, χρήματα για να προωθούν για να λένε στους ανθρώπους ελάτε στην Ευρώπη και από την άλλη πλευρά να τους λέμε μην έρχεστε στην Ευρώπη. Κάποιος θα πρέπει να αποφασίσει τι θέλουμε να κάνουμε. Θα πρέπει να τα εξισορροπήσουμε όλα αυτά. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για τα θέματα ασφάλειας αλλά θα πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά με, έναν έξυπνο τρόπο χωρίς να σκοτώνουμε την οικονομία. Αυτή είναι μία πρόκληση. Ασφάλεια από τη μία πλευρά ε, και φιλικότητα από την άλλη. Κύριε Πρόεδρε, αυτές είναι μερικές από τις προκλήσεις με τις οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωποι για μία ακόμα φορά. Στρεφόμαστε σε εσά και ε, παράλληλα σας ευχαριστώ για το ότι μου δώσατε το λόγο, τον οποίο καταχράστηκα φαντάζομαι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. for Σας ευχαριστώ κύριε Ριφάη για την καταπληκτική σας ομιλία. Ακολουθεί συζήτηση. Ο Ιστφαν η πρώτος που είναι πρόεδρος της ειδική ομάδας του τουρισμού και αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας, η οποία διοργάνωσε και την επίσκεψή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στη γλώσσα μου. Γι' αυτό βάλτε τα ακουστικά σας. Ευχαριστώ πολύ. Από χθε βρίσκομαι δίπλα στο Γενικό Γραμματέα και κοιτάω τα διάφορα προγράμματα και πραγματικά δεν ούτε στιγμή. Πραγματικά ήταν καταπληκτικά τα όσα μας είπε για τον τουρισμό. Για εκείνον δεν είναι μια βιομηχανία όπως οι άλλοι, δεν είναι τεχνικά θέματα. Είναι ένας τρόπος για να βλέπει τον κόσμο. Θέλει να χρησιμοποιηθεί ο τουρισμός για να δημιουργηθεί μια καλύτερη ζωή για πολλούς ανθρώπους. Μας μίλησε για πολλά προγράμματα και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Γενικό Γραμματέα που δέχτηκε την ε, πρόσκλησή μας. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ε, ανέλαβε το τομέα του τουρισμού, αλλά η πρώτη φορά που έρχεται να μας επισκεφτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω να μην είναι η τελευταία φορά, γιατί σήμερα θα ήθελα να προτείνω μία πρωτοβουλία και ελπίζω να τύχω τη υποστήριξή σας. Νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από τον Μάντι Σούλ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να συνάψει μία συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανώσεων, γιατί υπάρχουν παρεφερείς συμφωνίες με άλλες οργανώσεις, δεν υπάρχει όμως μια συμφωνία με εμάς, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ορισμένοι θεωρούν ότι ο τουρισμός δεν είναι και τόσο σημαντικός. Αρκεί το να έχει κανείς νομοθεσία. Η νομοθεσία όμως, λένε, δεν είναι αρκετή για τον τουρισμό. Μιλώντας στο Γενικό Γραμματέα και ακούγοντας ε, τις εξηγήσει του για το τι μπορούμε να πετύχουμε, πόσα μπορούμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, Νομίζω ότι εδώ στην Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο, θα πρέπει να δεχτούμε αυτή την πρόκληση. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να ενδυναμώσουμε τον ευρωπαϊκό τουρισμό έτσι ώστε να παίξει πιο καθοριστικό ρόλο στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Έχω την εντύπωση ότι εδώ στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο αυτό που ενδιαφέρει τους ανθρώπους είναι η δημιουργία προσκομμάτων στον τουρισμό. Προσπαθούν να, να, στο, να τον σπρώξουν στο βάθος της σκηνής. δεν θέλουν να βοηθήσουν τον τουρισμό. Είναι καταπληκτικό λοιπόν το ότι έχουμε εδώ μεσά μας το Γενικό Γραμματέα γιατί υπάρχουν συνάδελφοι εδώ που εκπροσωπούν τη βιομηχανία. Η βιομηχανία αναζητάει εταίρους σε μας. Αν θέλετε η Ευρώπη να συνεχίσει να είναι ο βασικός τουριστικός προορισμός, είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε. Η Επιτροπή μας, στην Επιτροπή μας θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο τουρισμός δημιουργεί θέσεις εργασίας και φέρνει επενδύσεις, φέρει πλούτο στην Ευρώπη. Και θα πρέπει πραγματικά να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Το τελευταίο 1,5 χρόνο βίωσα πολλές περιπτώσεις όπου εμπόδια και ε, υπήρξαν εμπόδια στον τουρισμό και όχι μία διευκόλυνσή του. Βεβαίως ε, οργανώνονται εξρατείες και μας, αυτό μας βοηθάει να προχωρήσουμε. Δεν θα πρέπει όμως να φύγουμε από εδώ και να σταματήσουμε τις προσπαθίες μας. Ευχαριστώ πολύ τον Γενικό Γραμματέα που ήρθε, ευχαριστώ τους συναδέλφους που έδωσαν τη στήριξή τους, την Κλάουντια για παράδειγμα, καθώς και όλους μου τους συναδέλφους που είναι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν τον τουριστικό κλάδο. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή την διαδικασία έτσι ώστε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των δύο οργανώσεων και ελπίζω να υπάρξει και υποστήριξη και από τη δική σας πλευρά. Εγώ θα ζητούσα από τους συναδέλφους μου να βοηθήσουν την επόμενη χρονιά και να μας υποστηρίξουν ως προς τις δράσεις που αναλαμβάνουμε σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πέτρο Όρτο που πραγματικά δραστηριοποιήθηκε στην Επιτροπή μας και τον Κάλλο Κροάστα από την ε, Γενική Διεύθυνση. Χθε είχαμε την ε, ε, ευκαιρία να τους ακούσουμε και υποσχεθήκαμε ότι την επόμενη χρονιά η Επιτροπή θα διαδραματίσει περισσότερο ενεργό ρόλο. Και θα ήθελα να δώσω του λόγο στου συναδέλφου, μου, αν κάποιο θέλει να μιλήσει. Ευχαριστώ. Ο Λουίς Δεγκράντε Πασκουάλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και καλωσορίσατε κύριε Ριφάη. Τα λόγια σας είναι ένα σύνολο ευχολογίου, καλών προθέσεων και μιας ανάλυσης που όλοι είμαστε σύμφωνοι αυτό από τη μια είναι καλό και από την άλλη είναι ανετικό. Ο πρόεδρος τα είπε πολύ καλά από την αρχή. Έχουμε ένα πλαίσιο δράσης που περιορίζεται από το άρθρο 195 της συνθήκης. Δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα, είναι ε, μάλλον δεύτερης κατηγορίας αρμοδιότητα και σύμφωνα με την επικουρικότητα βρίσκεται στα χέρια των κρατών μελών. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία αλλά είναι τόσο σημαντικός ο τουρισμός και τόσο ισχυρός που ξεπερνάει το πλαίσιο των ίδιων μας των κανόνων και των συνθήκων. Ξεχυλίζει δηλαδή και θα πρέπει να το σταματήσουμε το νερό αυτή την πλημμύρα. Και όταν υπάρχουν αξιέπαινες ε, πρωτοβουλίες, είναι καλές, αλλά θα πρέπει η ίδια Επιτροπή να έρχεται να μας ανακαλεί στην τάξη. Προσοχή, έχουμε νομικό πλαίσιο. Δεν μας επιτρέπονται πολλά πράγματα. Εγώ είμαι εδώ 11 χρόνια η Επιτροπή μας δεν έχει ξεχάσει ποτέ τον τουρισμό. Έχουμε ασχοληθεί από την πρώτη μέρα ορισμένοι από εμάς. Θα πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας ότι ο πλούτος του τουρισμού βγαίνει από τον ανταγωνισμό. Και τα κράτη μεταξύ αυτών και το δικό μου που έχουν ως βασικό κλάδο της οικονομίας τον τουρισμό και έχουμε σπάσει και το ρεκόρ στην ιστορία μας. Θέλουμε να ανταγωνιστούμε με τους άλλους, θέλουμε να συμμετέχουμε με τις δυνάμεις μας, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να υπάρχουν και ρυθμίσεις. Ο ίδιος ο κύριος Ριφάη μίλησε για σημαντικά ζητήματα, ε, μίλησε για τη Βαρκελόνη που είναι καλό παράδειγμα για το πώς ξεχυλίζει και υπερβαίνει ε, τους κανόνες. Έχουμε νέα συνεργατική οικονομία. Οι νέοι ταξιδεύουν, θέλουν να ταξιδεύουν και να μένουν σε φτηνά διαμερίσματα ας πούμε. Ε, δεν είναι καλό αυτό ή κακό, αλλά αυτοί που δυσανασχετούν είναι οι ξενοδόχοι, διότι πληρώνουν ε, φόρους και εμείς εδώ πέρα λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Mm. Και διαμαρτύρονται. Και μάλιστα τόσο πολύ ξεχυλίζει που η Κίνα που δεν είναι ακριβώς υπόδειγμα δημοκρατίας ε, εισβάλλει παντού στην Ευρώπη. Το είδατε πρόεδρε. Στη Μαδρίτη τουλάχιστον φαίνεται ε, και πηγαίνουν και απευθύνονται ε, στα μαγαζιά και όλοι στα κινέζικα στους πελάτες γιατί είναι οι τουρίστες που έχουν λεφτά είναι η κινέζικη μεσαία τάξη. Άρα ο τουρισμός είναι και ένας τρόπος εκδημοκρατισμού, ένας τρόπος να παγκοσμιοποιούνται οι αρχίες και οι αξίες και η Ευρώπη μπορεί να δώσει παράδειγμα εδώ ηγετικό. Στο μέλλον θα έχουμε μια ποσόστοση λέει 40% αλλά το είπε πολύ καλά κύριος Ριφάη αυτό θα είναι ακόμα πιο παγκόσμιο και πραγματικά μας έχει ξεφύγει το σύστημα. Δηλαδή 500, τόσο 560 εκατομμύρια τουριστών επισκέφτηκαν την Ευρώπη. Έχουμε κανόνες, πρέπει να τους στηρούμε, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχει αλλάξει η κατάσταση και με ένα έμεσο τρόπο θα πρέπει να σπάσουμε, να ξεχυλώσουμε αυτό το κορσέ που έχουμε βάλει οι ίδιοι στον εαυτό μας για να μπορέσουμε να τα διαδώσουμε όλα αυτά, τις αξίες, την οικονομία, τον πλούτο και τον πολιτισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Ταπαρδέλ. Ευχαριστώ. Κύριε Ριφάη, καλώς ορίσατε. Για μένα είναι τεράστια χαρά ότι σας συναντούμε. Διότι ο τουρισμός δεν έχει ξεχαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι κατά τη θητεία αυτήν στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Πολλοί συνάδελφοι ε, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα από όλες τις πολιτικές ομάδες για τον τουρισμό. Και αυτό με ικανοποιεί γιατί δημιουργήσαμε μία ειδική ομάδα Task Force με 140 βουλευτάς όλων των πολιτικών ομάδων σχεδόν και όλων των επιτροπών διότι ο τουρισμός σχετίζεται με πολλές επιτροπές, όχι μόνο μεταφορών και γι' αυτό μπορούν να γίνουν οριζόντιες συζητήσεις και με άλλες επιτροπές που αφορούν και αυτές τον τουρισμό. Ο λόγος σας με συγκίνησε διότι και εγώ ξέρω ότι ο τουρισμός χρειάζεται ανθρώπους που τον αγαπούν παθιασμένα και που ζουν γι' αυτόν και καταλαβαίνουν σε τι βαθμό είναι σημαντικός οικονομικά αλλά και κοινωνικά. Θα ήθελα τώρα να σας θέσω ένα πιο συγκεκριμένο ερώτημα γιατί προσπαθούμε και εμείς να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου για τη σημασία του τουρισμού στην Ένωση. Θα θέλαμε το 2018 να οριστεί Ευρωπαϊκό Έτος Τουρισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ξέρω ότι τα Ηνωμένα Έθνη επίσης μπορεί να ορίσουν ένα έτος για τουρισμό και βιώσιμη ανάπτυξη το 17. Και αυτό μας ικανοποιεί, με ικανοποιεί. Μπορείτε να μας πείτε τίποτα για αυτή την πρωτοβουλία. Επίσης, θα ήθελα την υποστήριξή σας για τη δική μας πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Έτους Τουρισμού είναι μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί από κοινού μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιών. Και φυσικά χρειάζεται υποστήριξη των χωρών μελών και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη θα ήταν πρόσδεκτη. Μιλήσατε για τις τρομοκρατικές επιθέσεις, για τα προβλήματα της ασφάλειας. Φυσικά εδώ αυτά έχουν επιπτώσει και στον τουρισμό, αλλά αναρωτιέμαι πώς θα μπορούσα με εμείς οι εκπρόσωποι των χωρών μελών που ασχολούμαστε και με προβλήματα άμυνας, πώς να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ο τουρισμός δεν είναι απόλυτα, δεν εξαρτάται απόλυτα με την ασφάλεια και τα προβλήματα ασφάλειας. Πώς να το εξηγήσουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα ως προς το καθεστώς απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Κάθε επίθεση έχει επιπτώσεις Οι συνάδελφοι διστάζουν όλο και περισσότερο και νομίζω ότι ο τουρισμός θα μπορούσε να τα μας ενώσει όλους και να δημιουργήσει πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ των λαών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, η Jill Thank you. Um, and thank you Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος σας ήταν ενδιαφέρον και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για μερικά από αυτά που είπατε για τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίω, διότι εκπροσωπώ την Ουαλία από το Ηνωμένο Βασίλειο και εκεί θα οργανωθεί σε λίγο δημοψήφισμα για την παραμονή μας στην Ένωση. Οι περισσότεροι Ουαλοί θέλουν να παραμείνουν στην Ένωση και γι' αυτό ετοιμάζουμε οικονομικά και πρακτικά επιχειρήματα και γι' αυτό μου άρεσαν τα παθιασμένα σας επιχειρήματα υπέρ της Ένωσης. Μας βοηθήσατε πολύ. Στην Ουαλία βλέπουμε, ξέρουμε τη σημασία του τουρισμού για την οικονομία μας. Το 2016 δε θα αρχίσει να χορηγείται ένα νέο δίπλωμα τουρισμού στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας διότι έχουμε πολύ ωραία χώρα ενδιαφέρουσα γλώσσα και πολιτισμό και θεωρούμε ότι και αυτό είναι τμήμα της βιωσιμότητας αναρωτιόμουν μήπως μπορούσατε να μας δώσετε κανένα παράδειγμα συνδυασμού κλιματολογικής, πολιτικής και προώθησης του τουρισμού. Και κάτι άλλο, πώς μπορούμε να εγγυηθούμε τα κοινωνικά συμφέροντα των υπαλλήλων. Θέλουμε να υπάρχουν δουλειές και θέσεις εργασίας καλής ποιότητας με αξιοπρεπείς απολαβές. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε ο Πέτερ Λούντγκριν. Ευχαριστώ πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Καλώς όρισατε κύριε Ριφάη. Όπως βλέπετε είναι πολύ διαφορετικές οι απόψεις που έχουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ την Ευρωπαϊκή Ένωση τη θεωρώ αποτυχία. Υποτίθεται ότι πρόκειται για ελευθερία, για ελεύθερη διακίνηση, για εμπόριο, για ελεύθερη κυκλοφορία. Και πού κατέληξε, πού κατάντησε σε ένα γραφειοκρατικό τέρας. Ε, και έχει και τις φιλοδοξίες να γίνει μεγάλη δύναμη. Μεγάλη αποτυχία ο τουρισμός μέχρι τώρα έχει ξεφύγει από τα νύχια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει παραμείνει σε εθνικό επίπεδο και κυρίως τοπικό επίπεδο. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη η οποία αποφασίζει για το που εγώ θέλω να πάω τουρισμό, να ταξιδέψω. Άκουσα τώρα για την Ουαλία Εγώ δεν ε, ταξιδεύω κάπου επειδή θα μου πει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τι ωραία που είναι και να πας εκεί διακοπές. Θα πάω εκεί που θέλω και στα μέρη που με ενδιαφέρουν. Ε, δεν θα μου πει κανείς που θα πάω διακοπές. Λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητο στοιχείο ε, και εταίρος για τον τουρισμό. Γιατί πιστεύετε ότι δεν μπορούν τα κρατη να τα κάνουν μόνα τους όλα αυτά. Δεν υπάρχουν και πολλά παραδείγματα χωρών ε, μάλλον υπάρχουν ε, χώρες πολύ τουριστικές, η ε, Ισπανία, η Ελλάδα, που μια χαρά τα καταφέρνουν μόνες τους. Τι θέλουν την Ένωση. Και σε αυτά τα μέρη εγώ πηγαίνω. Υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στην Ισπανία πας για τον ήλιο, ας πούμε. Στη δική μου χώρα, που είναι η Σουηδία, για τις μεγάλες εκτάσεις, την αχανή φύση, την ησυχία, τη σιωπή, τη σχέση που έχουμε με τη φύση. Ε, έχουμε ε, την ιδιαίτερη αυτή ε, σουηδική ζωή. Τι δουλειά έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακατεύεται σε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κλούν. I'll go this side, I think. <laughs> oh, this one is on, yeah. Okay, thank you very much, and thank you for the um, for your contribution. Most um, Ευχαριστώ πολύ. Συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ο τουρισμός ε, και στην Ευρώπη, αλλά και σε επίπεδο παγκόσμιο. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ε, πόσο μεγάλη πρόκληση μπορεί να είναι οι κλιματικές αλλαγές ε, για φτωχές κοινότητες των οποίων η εξάρτηση από τον τουρισμό είναι μεγάλη. Καταλαβαίνω βεβαίω την αξία που έχει ο τουρισμός από οικονομική άποψη, Οκτώ εκατομμύρια θέσεις αφορούν τον τουρισμό, το 6% του ΕΠ. Φανταστείτε τις περιοχές που είναι μακριά από τα αστικά κέντρα. Εμεί σκεφτόμαστε βασικά τα αστικά κέντρα, υπάρχουν και άλλες περιοχές που έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά στην Ευρώπη. Υπάρχουν ε, τουρίστες που τους ενδιαφέρει περισσότερο η φύση και νομίζω ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά στην Ευρώπη για να καλύψουμε και αυτέ, αυτό το κλάδο του τουρισμού. Η Natura δηλαδή έπαιξε ιδιαίτερα ενεργό ρόλο σε κοινότητες που εξαρτώνται από τον τουρισμό. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος ε, της οικονομίας που αφορά τον τουρισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την sharing economy, είναι εδώ και θα μείνει και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι ένα γεγονός που αφορά άτομα, καταναλωτές που παίρνουν αποφάσεις μόνοι τους. Πάροχοι στον των ε, ε, ε, υπηρεσιών μεταφοράς είτε στέγασης. Βεβαίως θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι, να σέβονται ορισμένες, ορισμένα προπετούμενα της νομοθεσίας. Όλα αυτά όμως αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση για μας. Δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε όλα και να κάνουμε μια προσπάθεια να εμποδίσουμε την ανάπτυξή τους. Αυτή είναι μια πρόκληση και θα πρέπει να την ε, αρπάξουμε, γιατί οι καταναλωτές σε κάθε περίπτωση θα κάνουν τις δικές τους επιλογές. Συμφωνώ με πολλά από τα σχόλιά σας. Κάνατε μία αναφορά στην ε, τροποκρατία. Έχουν γίνει πάρα πολλές ε, συζητήσεις για αυτό το θέμα και σε ό,τι αφορά το κλείσιμο των συνόρων. Ναι, για να μπορούμε να ελέγχουμε ποιος μπαίνει στην Ευρώπη. Ενδεχομένως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένας άλλος όρος, αντί να μιλάμε για κλείσιμο το σύνολο, τι να κάνουμε, να βάλουμε ένα μεγάλο τείχο που να μην μπορεί να περάσει κανείς. Αναρωτιέμαι ποιο είναι το μέλλον της, της Ευρώπης. Οι επισκέπτες βεβαίως, αυτοί που επισκέπτεται την Ευρώπη, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Αυτά ήταν τα σχολιά μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα ιδιαίτερα διαφωτιστικά μας είπατε και σχετικά με, την, με τις κοινέ εμπειρίες που θα μπορούσαμε να έχουμε και να τις ε, ε, ανταλλάξουμε όλα αυτά έχουν και το επιπρόσθετο πλεονέκτημα ότι υπάρχουν διαφορετικοί πολιτισμοί και ο τουρισμός δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν ανταλλαγέ. Κύριε Γενική Γραμματέα, θα πρέπει να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας και θα πρέπει να σας πω ότι με χαροποιεί ιδιαίτερα η παρουσία σας. Είχα το προνόμιο να σας γνωρίσω πριν από τρία χρόνια και πραγματικά με γοήτευσαν τα όσα είπατε. Είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου όταν εκλεγήκατε για τη δεύτερη θητεία σας. Στη συνάντηση αυτή τα παρούσες πάνω από 100 χώρες και όλοι ψήφισαν υπέρ ημών. Πραγματικά αυτό είναι άνευ προηγουμένου. Ο υποψήφιος δεν ήταν παρόν όταν έγινε η συζήτηση, αλλά Τώρα μπορώ να σας το πω, δεν είχα την ευκαιρία να το κάνω στο παρελθόν, σε όλες τις συζητήσει, όλες οι χώρες, οι παριστάμενες είπαν ότι ήσασταν ο τέλειος άνθρωπος σε αυτή τη θέση. Αυτό το βλέπω στην ε, ε, σημερινή σας ε, παρέμβαση. Ο κύριος Ριφάη βλέπει με πάθος τον τουρισμό. Μας χρειάζεται πληροφόρηση. Συμφωνώ μαζί σας. Θα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία με την Παγκόσμια Οργάνωση Τουρισμού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην ομάδα του κυρίου Ριφάιλ βρίσκονται και νέοι που γνώρισα όταν ήμουν υπουργό τουρισμού και θα πρέπει να σας πω ότι είναι άνθρωποι πραγματικά καταρτισμένοι. Η Παγκόσμια Οργάνωση Τουρισμού είναι ένα χρυσορυχείο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσα έχουν κάνει για να μπορέσει να εξελιχθεί ο τουρισμός στην Ευρώπη. Εγώ ήμουν εισηγήτρια για τα θέματα της εσωτερικής αγοράς αυτό αφορούσε ε, την προώθηση του τουρισμού, νέες μέθοδοι για την προώθηση του τουρισμού. Είναι σαφές, στην Ευρώπη υπάρχουν διαφορές. Εμείς όμως εδώ σε αυτή την έκθεση θα έχουμε τροπολογίες. Ε, υπήρξαν τροπολογίες οι οποίες ε, είχαν στόχο μία ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Παγκόσμιας Οργάνωσης του Τουρισμού. Αυτή, αυτό, αυτή η ανταλλαγή εμπειριών είναι ιδιαίτερα σημαντική για να μπορέσει να αναπτυχθεί αυτή η βιομηχανία που δεν είναι μία άκαμπτη, ξηρή βιομηχανία. Είναι μία βιομηχανία που μπορεί να προωθήσει, να, να συμβάλλει στην ειρήνη στον κόσμο. Όταν γνωρίζει κανείς τις παραδόσεις ενός τόπου, τις καταλαβαίνει καλύτερα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καδίας και να σας πω ότι εύχομαι η εμπειρία σας να μπορέσει να βοηθήσει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και ο πρόεδρός μας και τα μέλη αυτής της Επιτροπής δίχως άλλο θα μπορέσουν να πείσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών. Ένα τρίτο σημείο που αναφέρατε ότι δηλαδή θα πρέπει να παίξουμε ηγετικό ρόλο σε αυτό το τομέα. Οι μεταφορές είναι σαφές ότι στην έκθεση θελήσαμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σήμα. Είναι πολύ πιο εύκολο να προωθήσουμε την Ευρώπη ως χώρα προορισμού. Όταν ήμουν υπουργό στη Ρουμανία έλεγα ότι το σημαντικό δεν είναι οι ετικέτες. Το σημαντικό είναι να κοινοποιήσουμε αυτό το σήμα κατά τεθέν στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τις εμπορικές σχέσεις και τη ε, δυνατότητα ας πούμε ανάπτυξη περαιτέρω σχέσεων με την Κίνα. Γιατί δεν μπορεί να έχει κανείς ε, τουρισμό όταν δεν υπάρχουν ανταλλαγές. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα έχετε κάνει για την πρόθεση του τουρισμού στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Η Κλάουδια Μοντέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τουρισμού του ΟΗΕ για την προσέλευσή του. Δεν είναι πρώτη φορά που τον ακούω και πάντοτε οι λόγοι του είναι εμπνευσμένοι και γνωρίζει το αντικείμενό του. για το οποίο ενδιαφερόμαστε και τόσοι πολλοί από εμά όπως και εγώ. Η σημερινή του προσέλευση νομίζω ότι μπορεί να ξυπνήσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον της Επιτροπής μας στον τουρισμό. Τι να σας πω, τα είπατε όλα εσείς οι προηγούμενοι. Από την αρχή της θητείας θελήσαμε να προωθήσουμε τον τουρισμό. Ο τουρισμός προφανώς δεν είναι απλώς ένας οικονομικός τομέας αλλά συμβάλλει και στην αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών στον τρόπο ζωής και κατανάλωσης και κάτι που προωθεί την πολιτιστική ποικιλομορφία. Και αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν σεβόμαστε όλες τις χώρες μέλη ή ότι ή την πολυμορφία. Θέλουμε να όλοι μαζί να προωθήσουμε την βιομηχανία του τουρισμού στην ποικιλομορφία. του. εξάλλου έχουμε και το σύνθημα ενωμένη στην ποικιλομορφία. Είναι γνωστές οι θετικές επιπτώσεις που έχει ο τουρισμός στην απασχόληση και που σε μερικές χώρες θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν όμως και δύο-τρεις απορίες που έχω. Πρώτον, μιλάμε συνήθως για θεωρίες, για ευχαιολόγια, ώστε να παίξει, να γίνει πιο ανταγωνιστικός ο τομέας αυτός και θα υπήρχαν τρόποι αύξησης της ανταγωνιστικότητας του τομέα. Έχουμε μια έκθεση μπροστά μας που μιλάει για τις επιπτώσεις της λεγόμενης shared economy. Υπάρχει η ψηφιοποίηση που αυξάνεται συνεχώς και είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν όλο και περισσότερα πρότυπα επιχειρησιακά και ηλεκτρονικά, επίσης και στον τουρισμό. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά. Δύσκολα. Και πώς θα διασφαλίσουμε την συνύπαρξή τους με τις παραδοσιακές μορφές τουρισμού. Με τι δε τρόπο μπορεί ο η Παγκόσμια Οργάνωση Τουρισμού να αυξήσει τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθεσινά νέα λένε ότι οι θεωρήσεις και η σχετική γραφειοκρατία θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο στις Ηνωμένε Πολιτείε. την ίδια στιγμή που το Κοινοβούλιο συζητάει τα προβλήματα της, του Σέγγεν και την απλοποίηση των θεωρήσεων. Δύο εκθέσεις μας δε εδώ θα σχετίζονται και θα περάσουν σε λίγο χρόνο τι φρονείτε κι εσείς για τις θεωρήσεις, τι φρονείτε. Σας ευχαριστώ λοιπόν ξανά για την προσέλευσή σας και συνεχίστε έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή την τόσο σημαντική συνάντηση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο κύριος Ριφά είναι εδώ για να μας μιλήσει ένα θέμα που μας είναι ιδιαίτερα προσφυλές, δηλαδή την ανάπτυξη του τουρισμού ως ευρωπαϊκή πολιτική. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του συναδέλφου Ίσπαν σε ό,τι αφορά την ανάγκη για ένα κοινό πρωτόκολλο μεταξύ μας για να είμαστε περισσότερο δυνατοί σε όσα κάνουμε και μετά οι προθέσεις μας να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες δράσεις. Πιστεύω ότι ο τουρισμός πραγματικά είναι ένα στοιχείο δύναμης οικονομικής και όχι μόνον γιατί μας εμπλουτίζει και πολιτιστικά και μας βοηθάει να πλησιάσουμε τους λαούς. Από τη στιγμή που γνωριζόμαστε είναι πολύ πιο εύκολο να επιτύχουμε τους στόχους μας. Είναι και ένας ε, βασικός στόχος, ένας πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το να ευνοηθεί η οικονομική ανάπτυξη, η απασχόληση ιδιαίτερα στις πιο φτωχές, στις πιο απομακρυσμένες, στις πιο περιφερικές περιοχές. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει ένας κοινό παρονομαστής που αφορά την βιωσιμότητα που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την οικονομική πολιτική του τουρισμού. Με τι τρόπους το είπαν αρκετοί συνάδελφοι και όσοι συμφωνώ. Ψηφιοποίηση. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε κατά αποκλειστικότητα να βασιστούμε στις περιφερειακές πολιτικές. Μέσω με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να φτάσουμε από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη. Και αυτό γίνεται με το ψηφιακό σύστημα. Αυτό είναι πραγματικά κάτι αδιαφυσβήτητο. Παράλληλα, διαφυλάτοντας την ποιότητα, γιατί δεν μπορούμε να το δεχτούμε ο τουρισμός να μεταφραστεί σε έναν πόλεμο παροχής όλων και λιγότερων ε, υπηρεσιών. Πιστεύω ότι επειδή ένας από τους στόχους είναι ο συντονισμός των πολιτικών του τουρισμού, ένα από τα προβλήματα λοιπόν είναι ο κατακαιρματισμός των αρμοδιοτήτων. Εμείς έχουμε ένα σημαντικό αριθμό ατόμων που ασχολούνται με τον τουρισμό. Ε, σε επίπεδο τοπικό και σε επίπεδο ενωσιακό. Και αυτό αποδυναμώνει τη δράση που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε. Τέλος, η παρούσα κατάσταση. Δίχως άλλο, Πολλές φορές παίρνουμε εσπευσμένα αποφάσεις που μας υπαγορεύει ο φόβος. Αυτό είναι κάτι κατανοητό. Πιστεύω όμως ότι ο δρόμος για μία απλοποίηση των θεωρήσεων είναι ο δρόμος που θα επιτρέψει σε όλους μια καλύτερη προσφορά προς τους τουρίστες. Θα ήθελα να μου πείτε παρακαλώ με τι θα μπορούσαμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το Κοινοβούλιο στέλνει σαφέστατα μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και σε ό,τι αφορά την sharing economy, την ε, οικονομία διαμοιρασμού πόρων και περιουσιακών στοιχείων. Το θέμα δεν είναι το να γεννηθεί μια πραγματικότητα ή να κατασταλεί μια πραγματικότητα, αλλά να ρυθμιστεί αυτή η πραγματικότητα. Η sharing economy δεν θα πρέπει να δαιμονοποιείται θα πρέπει να ε, ε, τοποθετηθεί μέσα σε ένα πλαίσιο έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή βάση και κοινέ προϋποθέσεις ε, από τη στιγμή που η προσφορά είναι ίδια για τον τουρίστα. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ο Παύλ Τέλιτσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που καλέσατε το Γενικό Γραμματέα. Ναι, Και σας ευχαριστώ και για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Και για το γεγονός ότι μπήκατε και λίγο στο πολιτικό πεδίο και μ' αρέσει όταν άνθρωποι που έχουν τέτοιες θέσεις αντί δική σας το κάνουν εδώ στο κοινοβούλιο. Πρέπει να πω ότι έχω πολύ προσφυλή σε μνήμες ε, από τον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Επί κομμουνισμού ήταν ε, μία από τις αποστολές στο εξωτερικό και μπόρεσα να πάω στη Μαδρίτη και είχα πάει στην αποστολή αυτή με έναν πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών της χώρας μου που είχε κάτι άλλες δουλειές στη Μαδρίτη αλλά εγώ είχα πάει εκεί για τον οργανισμό σας. Ε, λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να, ε, λένε ορισμένοι, να, να κατέβεται σε αρμοδιότητες ε, κρατών μελών. Αυτό είναι μια μεμονημένη άποψη του κυρίου Λούντγκρέν. Οι περισσότεροι κατανοούν και εκτιμούν το γεγονός ότι ο τουρισμός στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζεται από πολλές πολιτικές δεν μπορούμε να το βλέπουμε έτσι ξεκομμένα, αλλά υπάρχει η προστασία των καταναλωτών, οι διάφορες ευκαιρίες που έχουμε σήμερα να αγοράζουμε τουριστικά προϊόντα στο διαδίκτυο, πώς προστατευόμαστε. Όλα αυτά έχουν να κάνουν, αρχίζουν από τις μεταφορές, επενδύσεις στα διευρωπαϊκά δίκτυα, διασύνδεση διαφόρων τρόπων μεταφορών και συγκοινωνιών. Όλα αυτά ε, είναι σημαντικά ζητήματα αναντικατάστατα. Η Ευρώπη βεβαίως και είναι ε, ελκυστική και πολλές από τις χώρες μας, αλλά θέλουμε να έχουμε περισσότερους τουρίστες από παντού και η Πράγα και η Τσεχική Δημοκρατία είναι πάρα πολύ ελκυστική και είμαι βεβαίως ότι οι άνθρωποι που κάνουν 10.000 χιλιόμετρα για να έρθουν στην Πράγα δεν θέλουν να μείνουν μόνο στην Τσεχία αλλά θέλουν να κάνουν και άλλο τουρισμό, φυσιολατρικό τουρισμό, βιομηχανικό. Είναι περίπλοκο το θέμα και έχει πολλές ψυχέ. Και αν δεν καταλάβουμε ε, αυτό το χαρακτήρα πάντα θα είμαστε χαμένοι για να το πω έτσι. Τώρα δεν θέλω να μπω σε ε, πολλά και αξιόλογα σημεία που είπαν πολλοί συνάδελφοι, αλλά θα μου άρεσε πάρα πολύ και θα εκτιμούσα αν ε, στην απάντησή σας και στα καταληκτικά σας σχόλια, βέβαια το κάνατε και στην εισαγωγή, ε, αναφερόσασταν στο εξή. Ποια είναι η τάση, ποια είναι η πολιτική, ποια είναι η δραστηριότητα, ποια είναι η προοπτική ε, ξαναλέω, για να ε, προσελκύσουμε τουρίστες στην Ευρώπη και τι θα πρέπει να ενισχύσουμε και τι ε, να ενδυναμώσουμε. Και τι κάνουν λάθος τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι πάει στραβά. Θα θέλατε να μας πείτε λίγο την αίσθησή σας, πόσο συντονισμένη πιστεύετε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνουμε εμείς στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Ξέρω ότι έχετε ομολόγους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκτός αυτού, εμείς τι κάνουμε. Πώς εκπροσωπούμεθα εκεί, πώς ε, συντονιζόμαστε, ποια είναι η δυνατότητα να δράσουμε από κοινού σε παγκόσμια φόρα και μεταξύ αυτών το δικό σας. Θα θέλατε περισσότερη ε, συνεργασία, συντονισμό, πιο θεσμικό ή θεωρείτε ότι είμαστε εντάξει. Ρωτώ, δεν σημαίνει ότι ε, το υποστηρίζω, απλώς επειδή ανταλλάσσουμε απόψει στα ε, πλαίσια της Επιτροπής θα ήταν πολύτιμη και η δική σας συνεισφορά. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σουίτσα. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Ριφάη για την προέλευσή του. Έχω εντυπωσιαστεί από όσα άκουσα. Θέλουμε να προωθήσουμε τον ευρωπαϊκό τουρισμό για να παραμείνει σε ηγετική θέση στον παγκόσμιο τουρισμό και στη νέα οικονομία sharing economy και στην ανταπόκριση για τις κλιματολογικές αλλαγές και για όλα. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο δίλημα. Είπατε ότι η ασφάλεια δεν πρέπει να μας εμποδίσει να ταξιδεύουμε, αλλά το γεγονός είναι ότι έχει γίνει πρόβλημα πια. Ε, και εγώ είμαι αισιόδοξη και πιστεύω ότι θα λυθεί, αλλά προς το παρόν είναι πρόβλημα για τον τουρισμό. Είπατε ότι ο τουρισμός αντιπροσωπεύει 10% του ΑΕΠ της Ευρώπης. Εγώ είμαι από την Κροατία όπου αντιπροσωπεύει 17% του ΑΕΠ και το Ντουμπρόβνικ στο Ντουμπρόβνικ που είναι η πόλη μου, ο τουρισμός αντιπροσωπεύει 100% του ΑΕΠ. Αν είναι κανείς από, από κάποιο τουριστικό προορισμό, ε, φοβάται γιατί εξαρτάται απολύτως από αυτόν η οικονομία και απαιτείται κάποια μεγαλύτερη διαφοροποίηση ίσως. Συμφωνώ ότι η Ευρώπη πρέπει να μιλήσει με ενιαία φωνή και σας ευχαριστώ που είπατε ότι χρειάζεται συνεργασία. Αλλά και η πολυμορφία είναι μέρος της, οικονομικής της Ευρώπης. Τώρα για τη Βαρκελόνη που είπαμε. Αυτοί δεν έχουν το πρόβλημά μας. Εμείς έχουμε το πρόβλημα της εποχικότητας. Έχετε καμία απάντηση για αυτό το πρόβλημα. Ξέρω ότι χρειάζονται νέες επενδύσεις, νέα περιεχόμενα, αλλά όποτε αρχίζουμε να κάνουμε κάτι καινούργιο όπως γήπεδα γκολφ, παραπονούνται οι πράσινοι. Κροάτες. Οι πράσινοι Κροάτες. Και είναι δύσκολο να κάνουμε κάτι καινούργιο λοιπόν και η εποχικότητα του τουρισμού μας είναι εμπόδιο. Έχετε καμία πρόταση. Η πολιτιστική κληρονομιά και ο τουρισμός δεν μπορούν να διαχωριστούν αλλά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα που είναι ο μαζικός τουρισμός από τη μία με τα κουρασγερόπλια και ο λεγόμενος υψηλός τουρισμός από την άλλη. Πώς να συνδυαστούν Έχω ερωτήσεις και άλλες, αλλά για να εξοικονομήσουμε λίγο χρόνο σταματάω εδώ και ελπίζω η Ευρώπη να συνεχίσει να είναι ηγέτης με γιώτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάκοφτσιτς δεν είναι μέλος της Επιτροπής μας, γι' αυτό δεν ξέρω το μικρό σας, αλλά κατ' εξαίρεση σας δίνουμε το λόγο. Ε, εντάξει, ε, τελευταίος και καταϊδρωμένος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ριφάη, ε, κύριε Γενική Γραμματέα που ήρθατε στη σε αυτή. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε με διαφορετικό κάπως τρόπο ε, το θέμα του ευρωπαϊκού τουρισμού ή του τουρισμού στην Ευρώπη. Φέτος το Μάιο ήρθατε στην Κροατία και σε μια περιφέρεια στην οποία ζω και μάλιστα στο παρελθόν ε, ήμουν και περιφερειάρχης. Ε, ο τουρισμός είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ίστρια που είναι λόγο περιφέρεια και ε, πολλοί κόσμος ζει από τον τουρισμό εκεί. Ο κύριος Λούντκρεν και εγώ έχουμε ένα κοινό. Είμαστε εύσομοι. Για όλα τα υπόλοιπα διαφωνούμε. Το μόνο που μας ενώνει είναι αυτό. Ο σωματότυπος Είμαι πεπισμένος ότι η ενίσχυση του τουρισμού με τρόπο θεσμικό θα βοηθήσει και θα αυξήσει και την ανταγωνιστικότητα στα κράτη-μέλη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν κάποιος ε, ξεκινάει από την Κίνα ή από τις Ηνωμένε Πολιτείες, ε, θα επισκεφτεί διάφορες χώρες, όπως είπε και ο κύριος Τέλιτσκα προηγουμένως. Και στα πλαίσια αυτού του ταξιδιού έχει πολύ μεγάλη σημασία ο καλός συντονισμός στην Ευρώπη. Όταν ήσασταν στην Κροατία μιλήσαμε για τη διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό τουρισμό, βέβαια αυτή δεν εγκρίθηκε, αλλά τουλάχιστον αρχίσαμε να συζητάμε για αυτά τα θέματα, για το πώς θα δημιουργήσουμε ε, μια ευρωπαϊκή αρχή τουρισμού που να είναι ένα συντονιστικό σώμα. Δεν θέλουμε ε, νέα ε, δομή, νέο οργανισμό γιατί εδώ στα θεσμικά όργανα δεν μιλάμε αρκετά για τον τουρισμό. Η κυρία Ντεμόντε έχει κάνει μια έκθεση εξαιρετική κατά τα άλλα, αλλά αυτό είναι το μόνο που έχει γίνει για τον τουρισμό τα τελευταία χρόνια. Ε, ο πρόεδρος της ειδικής ομάδας ε, τουρισμού είναι βέβαια πολύ ε, προσιλωμένος σε αυτή την προσπάθεια, αλλά είναι γεγονός ότι η Ευρώπη δεν είναι τόσο δημοφιλής προορισμός πριν από 10 χρόνια είχαμε 60% των ε, αφήξεων και τώρα είναι 50% και μετά μειούμενη 40% στο μέλλον των παγκοσμίων ε, αφήξεων δηλαδή. Δεν νομίζω ότι τα κράτη-μέλη μπορούν από μόνα τους να το αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Σήμερα η Κροατία μπορεί να μην ενδιαφέρεται γιατί έχει άλλες ε, φροντίδες και βάσανα και αναπτύσσεται ραγδαία ε, τουριστικά, δηλαδή πάει καλά ο τουρισμός, αλλά δεν είναι νησίδα η Κροατία, παρόλο που έχει πολλά νησιά. Θα πρέπει από κοινού να δράσουμε. Ευχαριστώ. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Γενικέ Γραμματεύ. Νομίζω ότι στο ίδιο μήκος κύματος κινούμαστε. Όπως είπαν και άλλοι, ο τουρισμός είναι ένας τομέας που μπορεί να δώσει ακόμη περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης στις προβλέψεις μας λέμε ότι εδώ μέσα σε δύο χρόνια μπορεί να δημιουργηθούν ακόμη 5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης από τον τουρισμό στην Ευρώπη με 100 δισεκατομμύρια προστιθέμενη αξία παραπάνω. Επίσης συμμεριζόμαστε την ανάλυση για τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Είναι σημαντικό να στηρίξουμε τις προσπάθειες της βιομηχανίας μας για να ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητά της. προσπαθώντας παράλληλα να βελτιώσουμε και τα περιεχόμενα για τα business και επίσης την sharing economy και την digital economy, την ψηφιακή οικονομία χωρίς να εμποδίζουμε την ε, άνθηση διαφόρων και διαφορετικών υπηρεσιών γιατί πάνω απ' όλα η ελευθερία, η ελευθερία. Με αναλογικότητα βέβαια όλα αυτά. Φυσικά συμμεριζόμαστε και το θέμα της βιωσιμότητας του τουρισμού και της αντιμετώπισης των κλιματολογικών αλλαγών. Η Κομισιόν και γενικότερα η Ένωση είναι στην προτεραιότητα. Και είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να συμφιλιώσουμε την ενίσχυση της αγωνιστικότητας του τουρισμού με ε, την κλιματική αλλαγή και την πρόκληση που συνιστά ε, αρχής γενομένης από την μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κυκλική οικονομία που είναι πάρα πολύ σημαντική και στρατηγική. Επίσης, ε, υπάρχει και το θέμα της διευκόλυνσης θεωρήσεων διαβατηρίων. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πέρσι την σχετική πρόταση. Και εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να συμφιλιώσουμε την ασφάλεια που είναι υψής σημασία με τη διευκόλυνση θεωρήσεων διαβατηρίων. Άρα, έχουμε πολύ καλή συνεργασία με το δικό σας οργανισμό. Ε, ελπίζω να συσφίξουμε τις σχέσεις μας και τη συνεργασία στο μέλλον. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ε, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας και ε, ο επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για τον Τουρισμό, ο κύριος Ούχελη. Θα ήθελα να πω ότι με ικανοποιεί ιδιαίτερα ότι όλο και περισσότεροι βουλευτές το καθιστούν σαφές ότι θα επιθυμούσαν τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων στον τομέα του τουρισμού. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας πω ότι μιλάμε για 17-18 εκατομμύρια ευρώ Και κάποιος μίλησε για ένα έμεσο ποσό 25 εκατομμυρίων. Μιλάμε για ανθρώπους που εργάζονται στη βιομηχανία του τουρισμού, Ευρωπαίοι πολίτες. Ακριβώς αυτό κάνουμε, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Προσπαθώ λοιπόν να δώσω, θα ήθελα να δώσω το λόγο για, σε άτομα από αυτή την ε, ε, αυτόν τον κλάδο. Έχει γίνει ένα μανιφέστο από εκπροσώπους αυτής της οργάνωσης. Αυτό το μανιφέστο προσυπεγράφει από τις, ε, τους εκπροσώπους αυτού του κλάδου και πιστεύω ότι είναι σημαντικό για μας που λαμβάνουμε τις αποφάσεις εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Εντουάρντο Σαντάντα να μας πει πώς θα ήθελε η βιομηχανία συνεργαστούν μαζί τους. Εντάξει, δεν το είχαμε κανονίσει αυτό και δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Κανονικά θα έπρεπε να είχαμε δει τελειώσει. Εντάξει, εντάξει, σας ζητώ συγγνώμη. Από ό,τι φαίνεται, η πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μάλλον οι άνθρωποι είναι απεσιόδοξοι γιατί εμείς δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Ο πρόεδρος λέει ότι δεν είχαμε προβλέψει ότι θα μιλήσει η βιομηχανία. Τι να, τι να κάνουμε, τα συζητάμε τα πράγματα μεταξύ μας και οι πρόσωποι της βιομηχανίας πάνε σπίτι τους. Νομίζω ότι αυτό ε, θα ήταν σκόπιμο να τους δώσουμε δύο λεπτά για να μιλήσουν. Ε, αν ο πρόεδρος θεωρεί ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν το είχαμε προγραμματίσει, τι να πω, πόκειται σε εκείνον. Εγώ το όμως δεν συμφωνώ. Ausschuss hier αλλά εδώ εμείς είμαστε Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού και κανονικά ομιλούν εδώ μόνο οι βουλευτές που εκπροσωπούνται. Έκανα μία εξαίρεση, πραγματικά κάτι εξαίρεση και εξαιρετικά σήμερα και έδωσα και το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι ήθιστε. Πάντα είναι πάγια διαδικασία. Καμιά φορά υπάρχουν εξαιρέσει, αλλά θα πρέπει να το έχουμε κανονίσει εκ των προτέρων και να το έχουμε συνεννοηθεί. Θα δώσω το λόγο τώρα στο Γενικό Γραμματέα για να κλείσει. Παρακαλώ. I think I have witnessed the operational Νομίζω ότι βλέπω άμεσα από πρώτο χέρι τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και νιώθω και ε, ε, λίγο σε δύσκολη θέση, γιατί ξέρω ότι θα τα σκόπιμο να ακούσουμε αυτή την παρέμβαση. Υπήρξαν 13 ομιλητές, μου αρέσει ο ρυθμός ε, 13 σε αντίθεση με το γενικότερο αίσθημα. Αλλά τι μεγάλη πρόκληση το να μπορέσω να απαντήσω σε όλα τα σχόλια και σε όλες τις παρατηρήσεις. Θα προσπαθήσω λοιπόν να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω α, με τον καλό φίλο από την Ισπανία. Η βάση μας εμάς είναι στη Μαδρίτη. Και το, και σε αυτή την εκχύληση, δηλαδή σε αυτή την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του ε, τουρισμού. Ε, αν με κατηγορείτε για ότι είμαι υπερβολικά αισιόδοξο, ναι, ίσως έχετε δίκιο. Εγώ πιστεύω ότι όταν ξεχυλίζει το νερό δημιουργούμε ενέργεια. Ε, το διοχετεύουμε κάπου αλλού, δεν το σταματάμε. Νομίζω ότι ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το θέμα του έτους 2013. Δίχως άλλο θα το υποστηρίξουμε αυτό. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θεωρήσει το 2017 το έτος του βιώσιμου τουρισμού για ανάπτυξη. Και νομίζω ότι το ένα θα συμπληρώσει το άλλο και θα τονίσει και το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Στην ίδια παρέμβαση αναφέρθηκε ότι το θέμα της ανοιχτής αυτής στάσης θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην ανάπτυξη του τουρισμού. Είπα ότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν επιπτώσεις μετά από κάθε κρίση σε επίπεδο ασφαλείας. Η πείρα μας δείχνει ότι υπάρχει πάντοτε μία ε, ένα αποτέλεσμα, αλλά η βιομηχανία του τουρισμού δεν παραδίδει τα όπλα. Την περασμένη εβδομάδα ήμουν στο Παρίσι Έφτασα μισή ώρα πριν τα τραγικά γεγονότα και είδα, είδα πραγματικά πως αντέδρασε ο κόσμος. Και τη δεύτερη μέρα με ενδιέφερε να μιλήσω με τους ε, ξενοδόχους και μου είπαν ότι είχαν πάρα πολλές ε, ακυρώσεις. Πριν από μερικές μέρες όμως ε, επικοινώνησα ξανά αλλά και όλα έχουν επανέρθει στην προτέρα κατάσταση. Η κυρία από την Ουαλία Συμφωνώ με το θέμα του τουρισμού περιπέτειας. Η κυρία από την Ουαλία το συνέδεσε και με το θέμα των κλιματικών αλλαγών. Επιτρέψτε μου να πω το εξή. Εμεί στην Παγκόσμια Οργάνωση Τουρισμού συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλά από αυτά τα προγράμματα. Επιτρέψτε μου να πω το εξή. Η ανάπτυξη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προ όφελος του υπεύθυνου τουρισμού, του βιώσιμου τουρισμού, η βιώσιμη ανάπτυξη, όχι μόνο για θέματα ε, κλιματικά. Ε, θα πρέπει να μας απασχολήσει και η οικονομική και η κοινωνική και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα υπάρχει ένα project το οποίο αφορά μικρομεσαία ξενοδοχεία. Συνήθως υπάρχουν ε, μεγάλες εταιρείες που βρίσκονται πίσω από τα ξενοδοχεία και καταρχάς θα πρέπει να υποστηρίζουμε τις σωστές πολιτικές. Αυτό το project όμως, ε, το οποίο συνεργαζόμαστε, ε, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας των μικρομεσαίων ε, ξενοδόχων κατά 17% και μετατρέπει την ενέργεια που καταναλώνει στο ξενοδοχείο σε ανανεώσιμη ε, ενέργεια. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το ελέγξαμε σε πέντε ευρωπαϊκές πόλεις. Και εδώ θα ήθελα να επανέλθω στο σημαντική παρέμβαση του κυρίου Λάμπεργκ. Δεν θέλω να εκφέρω άποψη για την αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Λούντρεν. Δεν ε, με φοβίζει η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που προσπάθησα να πω είναι ότι προσπάθησα να μιλήσω για ένα μοντέλο. Ένα μοντέλο στο οποίο θα μπορούσαμε να αναφερόμαστε και αναφέρομαι σε όλο τον κόσμο, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εμείς οι οραματιστές κοιτάμε, προσβλέπουμε σε ένα καλύτερο ε, κόσμο ασφαλή, με εκτά σύνορα και ελεύθερο, ελεύθερο με ελευθερία λόγου και έκφρασης. Αυτό είναι το μοντέλο που με ενδιαφέρει. Συμφωνώ μαζί σας σε αντίθεση με αυτό που είπατε, ε, ότι ε, την πορεία θα τη χαράξετε εσείς, ε, που δεν, δεν είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αρχίσει να προωθεί συγκεκριμένου τόπους προορισμού. Ο προορισμός μπορεί να αφορά μία πόλη, μπορεί να αφορά ένα μουσείο, ένα αρχαιολογικό χώρο, δεν αφορά κατά ανάγκη μία χώρα. Αυτό είναι ευθύνη του προορισμού, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε να πω τρία πράγματα. Να πιστέψετε στη δύναμη αυτής της βιομηχανίας, γιατί η πολιτική βούληση ε, ε, καθιστά τα πράγματα ευκολότερα. Αν συνεχίζετε να το αντιμετωπίζετε ως ε, ένα θέμα δευτερεύουσας σημασίας, δεν θα αποδώσει ποτέ, δεν θα γίνει σημαντικό για το όλο τον κόσμο. Δεύτερον, φροντίστε έτσι ώστε να υπάρξουν πρότυπα και κανονισμοί να υπάρχει ένα πλαίσιο με το οποίο θα μπορεί να συμμορφωθεί κανείς. Και αν αυτό το ονομάζεται εξουσία κύριε ε, Λούγκριν, ναι, συμφωνώ. Τρία, θα πρέπει να μας βοηθήσετε να υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση ε, του θέματος του, του, του, ή και ευαισθητοποίηση για το θέμα του τουρισμού ο τουρισμός είναι ένας τομέας τόσο σημαντικός αλλά που δεν λαμβάνεται πρακώς υπόψη από τους Ευρωπαίους πολιτικούς και αυτή η τάση θα πρέπει να αντιστραφεί. Ο τουρισμός είναι πολύ πιο σημαντικός στις Μαλδίβες, στην Κούβα, στην Ινδονησία, στην Κίνα, στην Ιαπωνία τώρα, σε πολλά μέρη του κόσμου. Πολύ πιο σημαντικό σε επίπεδο πολιτικό από ότι είναι στην Ευρώπη. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να, να εκμεταλλευτούμε αυτό το ενεργητικό που έχουμε. Ε, τέθη το ερώτημα γιατί η Ευρώπη είναι τόσο σημαντική. Είναι σημαντική γιατί είναι το λίγνο του τουρισμού, γιατί είναι η χώρα που, ο τόπος που γεννήθηκε ο, ο, τουρισμός. Παραμένει όμως ένας χώρος που αφορά το, δημο, το τον ιδιωτικό χώρο. Δεν είναι κάτι που ε, το έχει αγκαλιάσει ο δημόσιος χώρος. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας, η τουριστική βιομηχανία απασχολεί 12 εκατομμύρια άτομα, τα περισσότερα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλια που κάνετε για την ποιότητα των εργασιών. Δεν έχουν πάρα πολύ καλή φήμη οι εργασίες στον κλάδο του τουρισμού, γιατί παρεκκλίνουν από τα διεθνή πρότυπα. Εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε έτσι ώστε ε, να υπάρχει μια να ξεχωρίζει η Ευρώπη σε αυτό το τομέα. Συγχωρήστε με, έχω προβλήματα να διαβάζω το γραφικό μου χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο σημείο που έθιξε η κυρία από την Κροατία. Αναφερθήκατε στο θέμα της εποχικότητας. Δίχως άλλο έχει σχέση με τις θέσεις εργασίας. Η εποχικότητα είναι μία νόσος, είναι μία πρόκληση. Γιατί όταν επενδύεται σε κάτι και καταλήγεται να ποδίδει μόνο το μισό χρόνο, είναι μία χαμένη επένδυση. Είναι πρόβλημα για, για όλους. Και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να διαφοροποιήσουμε το προϊόν και να αυξήσουμε την ε, συνειδητοποίηση αυτού του προϊόντος. Ε, το να πηγαίνει κανείς ε, στη θάλασσα θα έλεγα, τολμάω να πω, ότι είναι πιο ρομαντικό να το κάνει το χειμώνα. Υπάρχει το φιούμε, η οπατία. Οι Αυστροούγγροι πήγαιναν εκεί το χειμώνα, γιατί είναι ένα μέρος που το χαίρεται κανείς και το χειμώνα. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε στις χώρες όλη τη Μεσόγειο. Κύριε Πρόεδρε, συγχωρήστε με, γιατί ξέρω ότι δεν απάντησα σε πολλές από τις ερωτήσεις που έγιναν. Ήταν 13 και οι 13 ήταν υπέροχες ε, και δεν θα μπορούσα να απαντήσω σε όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτή, για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε. Είναι τιμή μου κύριε, κύριε Πρόεδρε ε, το να συνεργαστώ μαζί σας σε μια προσπάθεια εδραίωσης ε, των σχέσεων με σας και με την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ριφάη για την καταπληκτική θαυμάσια παρουσίασή σας και τις απαντήσεις σας. Ήταν πολύ γόνιμη συζήτηση και ελπίζω να μας ξανάρθετε το συντομότερο.